Hello everyone. Good afternoon. Καλησπέρα σε όλους σας. Έχετε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Δεδομένου η ψηφοφορία αύριο θα κρατήσει πολύ, η ανταλλαγή απόψεων με τους νέους Ευρωπαίους που προβλέπεται για τις 11 και 30 θα αρχίσει στις 11, νωρίτερα δηλαδή. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, τότε γκρίνατε η μυρίσια διάταξη με την τροποποίηση αυτή. Επίσης, να ξέρετε ότι έχει υποβληθεί έτοιμα από την κυρία Γκόλτινγκ. Σήμερα το απόγευμα η συζήτηση για την ένσταση όσον αφορά την ασθετημιπηρίδη, το σημείο 8, να προωθηθεί, γιατί δεν θα είναι εδώ όλοι οι αρμόδιοι. Φοβάμαι όμως ότι δεν γίνεται, γιατί προτεραιότητα δίνουμε σε εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις και έχουμε πολλές σήμερα το απόγευμα. Και έχουμε επίσης και προσκεκλημένο απ' έξω μια συγκεκριμένη στιγμή στη συνεδρίασή μας για την έκθεση του IPCC. Ποτέ δεν είχαμε πει ότι για τις ενστάσεις θα τις συζητάμε μόνον εφόσον όλοι όσοι συμμετέχουν στην ένσταση είναι παρόντες. Ένας φτάνει. Ακόμα όμως και αν αλλάζαμε την ώρα της συζήτησης αυτής, δεν θα είχαμε εδώ τους αρμόδιους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά προς ενημέρωσή σας, οπότε θα παραμείνει το σημείο αυτό ως έχει. Εντάξει, ωραία, με ευχαριστώ. Αύριο τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φιλοξενήσει μια διάσκεψη υψηλού επίπεδου. Πρόκειται για την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την καινοτομία στην καθημερινή μας ζωή, βελτιώνοντας την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων. Μια success story. Η συνεδρίαση αυτή θα λάβει χώρα εδώ, στο ημικύκλιο. Και θα συζητήσουμε για την ε, ιατρική πρόοδο, την πιο καθαρή ενέργεια, ε, μηχανική ψηλού επίπεδου, προγράμματα έρευνα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι θα δείξουμε ποια είναι τα αποτελέσματα που ήδη έχουμε πετύχει, αλλά θα είναι και μια ευκαιρία για του πολιτικού να συζητήσουν μεταξύ του και να ακουστούν νέε ιδέε για την έρευνα και την καινοτομία. Η συζήτηση θα γίνει με πολίτες, με προσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, χώρες μέλη, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κτλ. Ο πρόεδρος Ταγιάννη και ο επίτροπος Μούντας είναι οι αμφιτρίονες από κοινού, όπου βέβαια είναι προσκεκλημένοι όλα τα μέλη των Επιτροπών ΕΝΒΙ και όλοι οι ευρωβουλευτές γενικώ. Οι περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είσαστε όλοι προσκεκλημένοι λοιπόν και ευπρόσδεκτοι. Παρακαλώ να έρθετε. Για σήμερα έχουμε 20 γλώσσες διερμηνία και όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά είναι διαθέσιμα. Επίσης θα μεταδοθεί από το διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Τώρα συστάσεις των συντονιστών από τη συνεδρίασή μας στις 20 Νοεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρηθούν εγκεκριμένε. Έρχομαι τώρα στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις διοργανικές διαπραγματεύσεις για τα λοιπάσματα πρώτα απ' όλα. Ε, μπορώ με ικανοποίηση να σας πω ότι υπάρχει μια προσωρινή συμφωνία η οποία πετέφθη την προηγούμενη εβδομάδα, την Τρίτη, μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Θα θυμόσαστε ότι το κύριο ζήτημα ήταν τα όρια καδμίου που επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα λοιπάσματα. Θέμα για το οποίο έχουμε εμεί αποκλειστική αρμοδιότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα όριο 60 μιλιγκράμμ ανά κιλό πρέπει να τεθεί επιπλέον αυτή η ωριακή τιμή θα αναθεωρηθεί, θα μειωθεί παρετέρω 7, μέρες, ε, συγγνώμη, 7 χρόνια μετά από τη θέση σε ισχύ της ρύθμισης αυτής. Η ψηφοφορία τώρα για τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν ε, με αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής μας θα γίνει τον Ιανουάριο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια στην κυρία Καρδίνη, η οποία ήταν η συγκητριά μας για αυτό το φάκελο. Μπράβο κυρία Καρδίνη. Έρχομαι τώρα και στην πρώτη έκθεση που θα συζητήσουμε σήμερα και που είναι του κύριου Μπέλετ και πρόκειται για την ε, οδηγία όσον αφορά τη διασυνοριακή υγεία. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους σας. Πράγματι, η εφαρμογή της οδηγίας αυτής για την διασυνοριακή υγεία, έτσι αυτό είναι το σημερινό μας θέμα, πάνω σε αυτό έχω ετοιμάσει και εγώ σχέδιο έκθεσης, όπου προσπαθώ να αναλύσω την κατάσταση και να διορθώσω κάποιες αδυναμίες που υπάρχουν. Να κάνω συστάσεις δηλαδή, ώστε να βελτιωθεί. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ότι οργανώσαμε πολλές συνεδριάσεις με τους ενδιαφερόμενους και μάλιστα αναφέρονται και στο νομοθετικό δελτίο που συνοδεύει την έκθεση αυτή. Προσκαλέσαμε επίσης Πολλού στην ακρόαση που οργανώσαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριο στόχος τη οδηγία αυτή, λοιπόν είναι να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε υπηρεσίες ε, υγείας εκτός της χώρα τους. Γιατί πολλές φορές χρειάζονται περίθαλψη ή φάρμακα σε άλλη χώρα πλην της δικιάς τους όταν ταξιδεύουν. Είναι βέβαια ένα περίπλοκο θέμα νομικά, γιατί έχουμε μεν αυτή την οδηγία, από την άλλη μεριά έχουμε και τον αρχικό κανονισμό του 2004 που αναφέρεται στο συντονισμό της ε, κοινωνικής ε, ασφάλειας, πράγματα που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης λοιπόν αξιολογείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Έρχομαι λοιπόν και πάλι στην εφαρμογή της οδηγίας. Οι χώρες μέλη έπρεπε να σωματώσουν στην εθνική νομοθεσία την ε, ρύθμιση αυτή πριν από το 2010. Τώρα επιτέλους το έχουν κάνει όλες οι χώρες. Ο κύριος στόχος λοιπόν τώρα της οδηγίας και του σχεδίου εκθεσής μου είναι η κινητικότητα διασυνοριακά των ασθενών. Και ακόμα και αν η κινητικότητα των ασθενών είναι σε χαμηλό επίπεδο μεταξύ των χωρών μελών, για ορισμένες κατηγορίες ασθενών, ασθενών που υποφέρουν από σπάνιες ασθένειες ή για ασθενείς που ζουν σε διασυνοριακές ε, περιφέρειες, λόγω της γεωγραφικής εγκύτητας, ε, πηγαίνουν από την άλλη μεριά των συνόρων, γιατί πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι πιο εύκολο για αυτούς τους ασθενείς. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς που ζουν σε διασυνοριακές περιφόρειες να μπορούν να έχουν αυτή την ευκολία. Στόχος λοιπόν της οδηγίας αυτής είναι να διευκολύνει ακριβώς αυτή την φροντίδα από την άλλη μεριά των συνόρων. Το γνωρίζουμε και ήμασταν σε επαφή με φόρουμ Ευρωπαίων Ασθενών και το γνωρίζουμε από πολλές περιπτώσεις ότι υπάρχουν πολλές πρακτικές και διοικητικές δυσκολίες γι' αυτό. Και αυτό ακριβώς είναι που και εμείς προσπαθούμε να αξιολογήσουμε για να καταργήσουμε όσο γίνεται περισσότερα εμπόδια. Το πιο σημαντικό εμπόριο σήμερα για τους ασθενείς είναι, είναι τα συστήματα αποζημίωσης. Δεύτερον, η εκ των προτέρων άδεια για μια τέτοια παροχή υπηρεσιών. Σε μερικές περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό να έχει πάρει εκ των προτέρων την άδεια ο ασθενής. Τρίτον, διοικητικές υποχρεώσεις που είναι πολλές και βαριές διαδικασίες συχνά. Έπειτα, πώς θα πληρώσουν οι ασθενείς αυτοί. Θα πρέπει να πληρώνουν από πριν, θα πληρώσουν μετά. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά συστήματα τα οποία δημιουργούν μεγάλη σύγχυση. Και έτσι οι ασθενείς δυσκολεύονται να πάνε να ζητήσουν εξυπηρέτηση από την άλλη μεριά των συνόρων, ενώ δεν είναι αυτό που θέλουμε. Για να διευκολυνθεί λοιπόν η κατάσταση όσον αφορά του ασθενείς, η πληροφόρηση των ασθενών είναι ζωτική σημασία. Χάρη στην οδηγία αυτή υπάρχει ένα δίκτυο σημείων επαφής σε όλες τις χώρες μέλη. Και υπάρχουν σε όλες τις χώρες μέλη Πράγματι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έτσι λύνονται και όλα τα προβλήματα. Για να πετύχει οδηγία είναι ζωτική σημασία όχι μόνο για τους ασθενείς αλλά και για τους επαγγελματίες του κλάδου. Να είναι όλοι πολύ καλά ενημερωμένοι για την οδηγία αυτή, για το τι προβλέπει, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν ισχύει ακόμα. Υπάρχει σαφώς έλλειψη πληροφόρησης και συνδυτοποίησης των ασθενών για τους περιορισμούς, τους διοικητικούς και τους οικονομικούς, αλλά και για τις ευκαιρίες που δίνει από την άλλη αυτή η οδηγία. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να αλλάξουμε. Πολλοί ασθενείς δεν γνωρίζουν ακόμα ούτε καν ότι υπάρχουν αυτά τα εθνικά σημεία επαφής. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν που πρέπει να φροντίσουμε. Οι ασθενεί λοιπόν δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Αν ας πούμε υπάρχει υπερβολική καθυστέρηση που πρέπει να κατευθύνουν τη διαμαρτυρία τους ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν, ποια είναι η διάρκεια της διαδικασίας. Και όπως είπα πριν, δυσκολεύονται γιατί δεν γνωρίζουν καλά πώς θα αποζημιωθούν ή κατά πόσο και πώς πρέπει να πάρουν εκ των προτέρων άδεια. Αυτά είναι κάποια εμπόδια και δυσκολίες λοιπόν που θέλουμε να απαλείψουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γι' αυτό και επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα στοιχεία, σε αυτά τα εμπόδια από τη μία και την έλλειψη πληροφόρησης, ενημέρωσης και συνειδητοποίησης από πλευράς των ασθενών. Στην έκθεση σε αυτά επικεντρώμαστε. Τώρα, μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή είναι ότι υπάρχουν ακριβώς αυτά τα εθνικά δίκτυα αναφοράς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κυρίως για ασθενείς που υποφέρουν από σπάνιες ασθένειες. Κάπου 6 8% των Ευρωπαίων πολιτών είναι αντιμέτωποι ή υποφέρουν από τέτοιες σπάνιες ασθένειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας είναι ζωτική σημασία για τους ασθενείς αυτούς. Υπάρχουν 24 τέτοια εθνικά δίκτυα αναφοράς ήδη προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες με τις σπάνιες ασθένειες. Μιλάμε βέβαια για οι ειδικέ γνώσεις που χρειάζονται, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα 24 δίκτυα αναφοράς με 900 έως 1000 περίπου ειδικευμένε μονάδες, 300 νοσοκομεία ανά την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτά τα εδά να λειτουργούν με τρόπο που να διευκολύνεται η συνεργασία και να χρησιμοποιούνται ευκαιρίες που προσφέρουν αυτά τα δίκτυα όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Τώρα μια ακόμα παρατήρηση σε σχέση με το Brexit. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στα πλαίσια αυτών ε, των δικτύων αναφοράς και της ειδικευμένης περίθαλψης υπάρχουν πολλά νοσοκομεία, 40 περίπου, στο Ηνωμένο Βασίλειο που συμμετέχουν. Θα θέλαμε να συνεχιστεί η συνεργασία με τα νοσοκομεία αυτά και στο μέλλον και μετά το Brexit. Επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να αναφέρω ακόμα και την πτυχή της ηλεκτρονικής υγείας, e-health. Ξέρω ότι αυτό το θέμα το εξετάζουμε σε διαφορετική έκθεσή μας. Παρ' όλα αυτά συνδέεται άμεσα, όπως καταλαβαίνετε, με την διασυνεργειακή περίθαλψη, ακριβώς γιατί η ηλεκτρονική υγεία αποκτά και μεγαλύτερη σημασία. Πρόκειται για την διαλειτουργικότητα των δεδομένων των ασθενών από την άλλη μεριά των συνόρων, προκειμένου να υπάρχει εμπιστοσύνη και ασφάλεια όσον αφορά τα δεδομένα αυτά και να συνεχίζεται η προσφορά φροντίδας την άλλη μεριά των συνόρων. Οι δυνατότητες της ηλεκτρονικής υγείας είναι τεράστιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στόχος της οδηγίας αυτής είναι να μεγιστοποιήσει το δυναμικό που προσφέρει αυτή η ηλεκτρονική υγεία σε σεβόμενοι απόλυτα βεβαίως πάντα το απόρριτο των δεδομένων των ασθενών. Ναι, μεν μεταφορά δεδομένων από την άλλη μεριά των συνόρων, αλλά με σεβασμό. Μιλάμε για έρευνα, μιλάμε για ανταλλαγή δεδομένων έρευνας διασυνοριακά. Και τέλος, θέλω να αναφέρω ιδιαίτερα στην έκθεση αυτή, αν και το είπαμε και στην αρχή, την περιφερειακή ε, μεθοριακή συνεργασία που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους ασθενούς που ζουν σε τέτοιες παραμαθόριες ε, περιοχές. Επειδή από την άλλη μεριά των συνόρων μπορεί να έχουν πιο κοντά οι υπηρεσίες που χρειάζονται από ό,τι στην ίδια τους τη χώρα, οικονομικά ή πρακτικά τους εξυπηρετεί περισσότερο, πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση εκεί χωρίς εμπόδια. Σε τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή είναι πιο λογικό να πάει στην άλλη χώρα ο ασθενής παρά στη δικιά του για τέτοιους πρακτικούς λόγους. Η οδηγία αυτή, είπαμε, υπάρχει από τη μία. Ε, χρειάζεται ο συντονισμός, όπως είπαμε, με τον κανονισμό του 2004. Το ότι συνυπάρχουν και τα δύο, η οδηγία και ο κανονισμός δηλαδή, συγχρόνως, δεν θα λέγω ότι δημιουργείται ακριβώ σύγχυση, αλλά ότι είναι περίπλοκα τα πράγματα και για τους ασθενείς, αλλά και για τους πάροχους υπηρεσιών υγείας. ανάλογα με την περίπτωση κανείς προτιμάει την εφαρμογή της οδηγίας ή την εφαρμογή του κανονισμού. Και αυτό είναι που περιπλάκει τα πράγματα. Γι' αυτό και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από ό,τι καταλαβαίνω είναι εδώ εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι, θα έπρεπε να δούμε μήπως μπορούμε να συντονίσουμε καλύτερα ή ακόμα και να συγχωνεύσουμε αυτές τις δύο νομοθετικές πράξεις, έτσι ώστε να είναι λιγότερο περίπλοκα τα πράγματα για το προσωπικό υγείας και τους ασθενείς. Είμαι ανοιχτό πάντως στις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των συναδέρφων που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπέλετ για την εισήγηση αυτή για την έκθεσή σας και τώρα να ακούσουμε τους κοιόδους εισηγητές, ο κύριος Βόλκε πρώτος. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για την κατά τη γνώμη πολύ πετυχημένη έκθεση και να πω ότι προσβλέπω στην καλή συνεργασία και χαίρομαι που μπορώ να πω ότι και οι δύο ενδιαφερόμαστε για την προστασία των δικαιωμάτων των ε, Ευρωπαίων ασθενών. Στόχος μας είναι να βελτιωθεί η διασυνοριακή περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διευκολύνουμε και τις επαφές ε, με τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων ε, στα άλλα κράτη-μέλη. Έχουμε το διασυνοριακό μέσο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί απολύτως όμαλα η διασυνοριακή περίθαλψη. Και ενώ η προθεσμία για εφαρμογή της οδηγίας έλεγε το 2013 είχαμε 26 διαδικασίες επί παραβάση. Πρέπει λοιπόν να ε, διευκολύνουμε τους ε, ασθενείς ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αυτή. με εκπλήσει το γεγονός ότι πολύ λίγοι ασθενείς γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος. Το Ευρωβαρόμετρο διαπίστωσε ότι μόλις το 20% των ασθενών το γνωρίζουν αυτό. Πιστεύω ότι είναι καθήκον μας να αυξήσουμε το ποσοστό αυτό. Όπως είπε ο εισηγητής, ε, σημαντικό ρόλο να παίξουν ε, έχουν τα σημεία επαφής. Ε, παίζουν ήδη σημαντικό ρόλο, αλλά οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν την δυνατότητα αυτή. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες προς τους πολίτες και να οργανώσουμε εκστρατείες πληροφόρησης. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να έχουν πληροφορίες οι πολίτες σχετικά με το τι δικαιούνται και τι όχι και να διευκολύνουμε τις διασυνοριακές διαδικασίες πληρωμών. Στην ψηφιακή ετούτη εποχή είναι απολύτως απαραίτητο αυτό και θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι έχουν σημαντικές και καλές δυνατότητες οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της υγείας. Προέρχομαι από κράτος μέλος όπου ακόμη οι συνταγές γιατρών δεν δίνονται ηλεκτρονικά, δίνονται ακόμη σε χαρτί. Τέλος, υπάρχει το θέμα της ε, συμβατότητα οδηγία και κανονισμού. Νομίζω ότι μπορούμε να το λύσουμε αυτό και προσλέπω στην καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρίης. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω σε αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, γιατί θέλω να ξεκινήσω από ένα νούμερο, πολύ απλό. Πέρυσι μόνο 203.000 αιτήσει αποζημίωση υποβλήθηκαν στις χώρες μέλη για ιατρικές πράξεις οι οποίες έλαβαν χώρα σε διαφορετική χώρα από τη δικιά τους πέρυσι, αλλά φαίνεται ότι είναι το ίδιο νούμερο λίγο πολύ τα τρία τελευταία χρόνια. 230.000 0,004% περίπου των συνολικών δαπανών των ιατρικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα είπε ο Ιβο Μπελέτη στην αρχή ότι υπήρχαν πολλές προσδοκίες από τους συναδέρφους όταν ψηφίσαμε την οδηγία αυτή για τη διασυνοριακή υγεία τον Ιανουάριο του 2011, θέλαμε κυρίως την ελευθερία για τον καθένα να μπορεί πρώτον να επιλέξει και δεύτερον να εξυπηρετηθεί με περίθαλψη και υπηρεσίε υγεία εκεί όπου προτιμά, είτε γιατί είναι πιο κοντά στο σπίτι του ή γιατί η κατάσταση τη υγεία του είναι τέτοια που χρειάζεται κάποια δίκευση που μπορεί να μην υπάρχει στη δικιά του χώρα. Θέλαμε επίσης αντιμετώπιση και διαδικασίες απλοποιημένες, λιγότερη γραφειοκρατία. Θέλαμε επίσης οι ασθενείς να μπορούν να προσφύγουν αν υπήρχε άρνηση εξυπηρέτησής τους και να έχουν όλη τη δυνατότητα εύκολα να έχουν ένα αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου και να μπορούν να τον πάρουν όπου θέλουν ε, μαζί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει οδηγία, ναι. Τα νούμερα όμως δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας. Οπότε πρέπει να ξέρουμε γιατί. Ο Ιβο Μπελέτ το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ψήφισμα εδώ με το οποίο ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει περισσότερα για την ψηφιακή μετατροπή της υγείας για το e-health, δηλαδή την ηλεκτρονική υγεία, με στόχο να είναι ο ασθενής στην καρδιά των αποφάσεων που τον αφορούν. Άρα, τα έχουμε όλα αυτά, έχουμε τη θεωρία, ε, δεν ξέρω αν έχουμε και το πνεύμα. Ε, τα εθνικά σημεία επαφής τώρα. Ποιος τα γνωρίζει, ποιος ασθενής γνωρίζει ότι υπάρχουν 10% μόνο των Ευρωπαίων έχουν ακούσει κάτι γι' αυτό. Αυτά λέει το Ευρωβαρόμετρο. Άρα δεν φτάνει να δημιουργηθούν αυτά τα σημεία επαφή, θα πρέπει και οι χώρες μέλη να τους δίνουν ε, τα μέσα που χρειάζονται για να λειτουργήσουν, να τα γνωστοποιήσουν στον κόσμο, να βοηθούν τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την τοπική γλώσσα επίσης. Υπάρχουν και άλλα εμπόδια, τα κριτήρια αποζημίωση, που είναι διαφορετικά μεταξύ των διαφορετικών χωρών μελών. Η γραφειοκρατία και πάλι, ε, η αναγνώριση των, της συνταγογράφησης Εντάξει, δεν λέω ότι είναι μαύρη εικόνα. Η οδηγία αυτή φυσικά και θα φέρει σημαντικές βελτιώσεις για τους ασθενείς. Υπάρχουν και τα νέα δίκτυα αναφοράς που συνδέουν τους ειδικού για τις σπάνιες ασθένειες. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τους συνδέει από ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα είναι η ιατρική γνώση που ταξιδεύει και να μην χρειάζεται ο ασθενής να ταξιδέψει απαραίτητα. Όλα αυτά δημιουργούν νέα δικαιώματα τα οποία δεν θα είναι χρήσιμα παρά μόνο αν τα γνωρίζει και ο πολίτης και ο ασθενής. Οπότε στηρίζω την έκθεση του συναδέρφου και ε, καλό θα ήταν να συντονιστούμε κάπως καλύτερα από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πεντιτσίνη. Όχι, δεν θέλει τώρα. Ωραία, άρα τελειώσαμε τους σκιώδεις εισηγητές που είναι εδώ παρόντες τουλάχιστον. Ποιος άλλος θέλει το λόγο? Ο κύριος Πέτερλε πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που ο εισηγητής πρόσεξε ιδιαίτερα το θέμα που επικρότησαν ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι ασθενείς στα κράτη-μέλη τους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ολοκληρωμένη προσέγγιση όπου πιστεύω ότι λαμβάνονται παρκώς υπόψη όλες οι κατηγορίες ενδιαφερομένων. Κάποιοι από εσά γνωρίζουν ότι υπήρξα ασθενής με καρκίνο και ξέρω πώς είναι όταν ένας γιατρός λέει ότι δεν μπορώ να σας βοηθήσω άλλο. Μπορεί να ζήσετε δύο, τρεις, τέσσερις μήνες ακόμη, αλλά αυτό είναι. Ξέρω περιπτώσεις από τη χώρα μου, όπου κατάφεραν να ζήσουν αρκετά χρόνια παραπάνω οι ασθενείς με καρκίνο, διότι είχαν επιτυχή θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος, σε άλλη χώρα μάλλον. Και αυτό δείχνει μια Ευρώπη που λειτουργεί καλά. Γνωρίζετε τι ευγνωμοσύνη νιώθουμε για κάθε παραπάνω μέρα ζωής που μας δίδεται και γνωρίζετε επίσης ότι αυξάνεται ο αριθμός των καρκινοπαθών. Χαίρομαι που βλέπω αυξημένη κινητικότητα. Δεν χαίρομαι όμως με τα χαμηλά επίπεδα κινητικότητας που υπάρχουν, όπως είπε και ο Ιβο Μπέλετ. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλύτερη οργάνωση για να βελτιώσουμε το σύστημα. Δεν θα επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν σχετικά με την ενημέρωση, με το δικαίωμα πληροφόρησης κλπ. Θα ήθελα όμως να θίξω όχι για πρώτη φορά το εξή. Η κινητικότητα των ασθενών έχει οδηγήσει και σε καλύτερη ε, διάδοση των γιατρικών γνώσεων, διότι θέλουμε να δούμε αυξημένη κινητικότητα και όσον αφορά τη γνώση. Θέλουμε δηλαδή ε, να διευρυνθούν τα δίκτυα των κέντρων αριστείας και Χαίρομαι που αναφέρθηκε το δίκτυο αναφοράς, διότι δεν υπάρχει ε, κάποιο μεμονωμένο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο το θέμα αυτό. Μόνο ως Ευρώπη μπορούμε να πετύχουμε προστιθέμενη αξία. Ιδιαίτερα, χάρηκα που ο εισηγητής αναφέρθηκε στις παραμεθόριες περιοχές. Αν είναι υπερβολικό το διοικητικό άχθος, Ε, τότε μπορεί να προτιμήσουν οι άνθρωποι να ε, ε, μετακινηθούν πολλά χιλιόμετρα αντί να περάσουν τα σύνορα και να διανύσουν πολύ μικρότερη απόσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σιερπέρεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, και ευχαριστώ τον Ιβο Μπελέτ το συζητήσαμε αυτό το θέμα με τον ε, Ιβο Πελέτ ε, και με τις ενώσεις ασθενών στην Ορλανδία. Σίγουρα και από το Υπουργείο και από τη Βουλή είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να έχει κανείς εξυπηρέτηση για την υγεία του από την των συνόρων. Έχουν γίνει βήματα έχει γίνει το πρώτο βήμα, αλλά ποιο είναι το δεύτερο βήμα τώρα. Ο κόσμος με σπάνιες ασθένειες, τι θα κάνει. Και αν δούμε τι έχει γίνει τον τελευταίο καιρό από την φαρμακευτική βιομηχανία, συχνά οι μέτοχοι αποφασίζουν τι θα πληρώσουν και τι δεν θα πληρώσουν και τι φάρμακα θα έχουμε και τι όχι. Οπότε εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει τα φάρμακα να είναι διαθέσιμα. Τι κάνουν όμως οι ασφαλιστές και τι κάνει η φαρμακευτική βιομηχανία. Υπάρχουν οι δυνατότητες, αλλά δεν είναι το μόνο εμπόδιο τα σύνορα. Και θα ήθελα στο κείμενο να μπει και κάτι πρέπει ο καθένας να μπορεί να έχει πρόσβαση. Εγώ καταλαβαίνω τα προβλήματα, ξέρω και με την ε, Ρωμανία το είχαμε συζητήσει για την ε, αντίσταση στα αντιβιωτικά. Σε άλλες χώρες προχωράν τα πράγματα, σε άλλες χώρες όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί. Οι χώρες μέλη όμως έχει μεγάλη σημασία το πώς αντιμετωπίζουν το θέμα. Όλοι κοιτούν, τώρα θα έχουμε και τις ευρωεκλογέ, όλοι ρωτάνε πού είναι η Ευρώπη. Να λοιπόν κάποια θέματα, και εδώ στρέφομαι προς τον Ιβο Μπελέτ, να θέματα τα οποία αγγίζουν τον πολίτη. Αν θέλουμε να είμαστε κοντά στον πολίτη, αυτό πρέπει να κοιτάξουμε, γιατί εκεί είναι που τον οι άνθρωποι και οι νέοι κυρίως πού είναι η Ευρώπη σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much. And now, uh, if there is no one else to take the floor. Ο κάποιον άλλον να ζητάει το λόγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ρίσου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στη συνεδρίασή σα. Ευχαριστώ τον εισηγητή τον κύριο Μπέλετ και τους κοιόδης εισηγητέ για την εξαιρετική τους έκθεση και για μια σειρά από θέματα που έχουν θέσει. Στον τρόπο και τη φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζουμε το όλο θέμα. Το πρώτο, όπως τα ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε έκθεση που απαιτείται από την οδηγία. Δημοσιεύτηκε κιόλα στις 21 Σεπτεμβρίου και στην έκθεση αυτή αναλύονται κάποια θέματα από αυτά που αναφέρει και η δική σας η έκθεση. Θα αναφέρω ορισμένα από αυτά. Η πρώτη οδηγία προσπάθησε να αποσαφηνίσει και να εγγυηθεί τα δικαιώματα των ασθενών διασυνοριακώς. Αυτό είναι μια από τι βασικέ μέρημνε της όλης νομοθετική μας προσπάθειας για να βεβαιωθούμε ότι τα δικαιώματα που απαιτούνται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ρυθμίζονται μέσα από αυτήν την οδηγία. Βέβαια, προέκυψαν και άλλε υποθέσει που εκδικάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οπότε χρειάστηκε να καλύψουμε και αυτέ. Η κινητικότητα φαίνεται ότι κάπω έχει αυξητική τάση αλλά όπως λέγεται και στην έκθεση, δεν υπάρχει και φοβερά δυναμικός χαρακτήρας. Η διασυνοριακή κινητικότητα των ασθενών δεν έχει αλλάξει το αντίκτυπο στον προπολογισμό των εθνικών συστημάτων υγειονομική περίθαλψης. Αυτό είναι σημαντικό γιατί στι συζητήσει που είχαμε κατά τη διαπραγμάτευση αυτής τη οδηγία ήταν ένα από τα βασικά νομοθετικά προβλήματα και φραγμού. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας με τα κάτι μέλη για να βελτιωθεί το επίπεδο τήρησης των κανόνων και να ευαισθητοποιηθούν και οι εθνικοί φορείς. Ένα άλλο θέμα που έχει ο εισηγητή είναι οι σχέσεις μεταξύ οδηγίας και των κανονισμών ε, κοινωνικής πρόνοιας σε εθνικό επίπεδο. Κάθε χρόνο πολλοί Ευρωπαίοι ε, πραγματοποιούν μικρότερα ή μεγαλύτερα ταξίδια στο εξωτερικό για λόγους υγείας αλλά εμποδίζεται η πρόσβασή του στο υγειονομικό σύστημα της άλλης χώρας λόγω των κανόνων. Ταυτόχρονα η οδηγία επικεντρώνεται στην αγωγή και τη φροντίδα. Αυτό δημιουργεί σύγχυση στους πολίτες, αλλά προσπαθούμε μαζί με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, την DG Sante, να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα πλέον και τις σχετικέ πληροφορίε θα τις λάβουν και τα σημεία επαφής καθώς και οι πολίτε κατ' επέκταση. Μια άλλη σημαντική προσπάθεια που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ο έλεγχο μεταφορά και συμμόρφωση. Όπω αναφέρθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε. ...26 διαδικασίες επί παραβάση λόγω της πλημελούς ή καθυστερημένης μεταφοράς. Όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και έχει κλείσει το σχετικό θέμα. Έχουν βγει και αποφάσεις. Τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση. Έλεγχος ε, συμβατότητας. Για να δούμε πώς εφαρμόστηκε, πώς υλοποιήθηκε στα εθνικά συστήματα η οδηγία με τις απαιτήσει της. Βεβαίως η οδηγία μπορεί να μεταφερθεί στα μέτρα και τα σταθμά των ε, εθνικών συστημάτων υγείας. Οπότε αυτό που κοιτάζουμε είναι πώς έγινε η υλοποίηση και πώς επηρεάζει τους πολίτες, αν υπάρχει διαφάνεια, πώς λειτουργεί το σύστημα. Το πρώτο θέμα που μας απασχολεί είναι η επιστροφή των εξόδων στην περίπτωση διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψης. Μετά η αδιαφανής τιμολόγηση και η άδικη μεταχείριση από ε, άλλα κράτη. Τρίτον, η προέγκριση της απαιτούμενης αγωγή και το περίπλοκο της όλης διαδικασίας και μετά ε, οι διοικητικέ διαδικασίε για να λάβει κανεί επιστροφή των εξόδων και βάσει τη προέγκριση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πετύχει ε, χειροπιαστά αποτελέσματα. Πολλά κράτη-μέλη αποφάσισαν να αλλάξουν την νομοθεσία του προ όφελο των ασθενών βάσει των όσων προέκυψαν και από το διάλογο που είχαμε μαζί του. Επόμενη, το επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχίσει τον εντατικό διάλογο με τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πιέσει για την σωστή μεταφορά τη οδηγία. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που έγινε η έκθεση και το είπαν και οι σχεδόν εισηγητές, είναι η έλλειψη ενημέρωση. Εμένει το πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό συνεχίζουμε τη δουλειά μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια σειρά από δράσεις, όπως εργαστήρια και σεμινάρια, αυτό που οργανώσαμε τον Οκτώβριο του 2016, παραδείγματι, για να συζητήσουμε με τους ενδιαφερομένους τα κράτη-μέλη, τα εθνικά σημεία επαφή, τι ενώσει ασθενών, πώ μπορούμε να ενημερώνουμε καλύτερα για τα δικαιώματά του του ανθρώπου. Επίση, αυτό μα έδωσε καλύτερο. Ετοίμασε το έδαφο για να συζητήσουμε με του ενδιαφερομένους και να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων πρόσφατα η εκστρατεία EUNME, e, η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ, που είχε στόχο κυρίω του νέου, με ενημέρωσε για προγράμματα ε, άτυπη και επίσημη υγειονομική περίθαλψη διασυνοριακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια προσπάθεια που την συνεχίζουμε σε συνεργασία με τα εθνικά σημεία επαφή και του βοηθούμε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, πιο αποδοτικοί, να βοηθούν του αισθανεί του και να τηρούνται οι κανόνε τη οδηγία. Γι' αυτό συναντιόμαστε συχνά μαζί τους Και έχουμε δώσει και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την ε, δράση των σημείων επαφής. 15 Νοεμβρίου μάλιστα εκδόθηκαν και αυτό ε, συνάδει πλήρω με, το με τόσα 16 της εκθεσής, της εκθεσής σας εδώ. Ε, η διασυνοριακή συνεργασία βλέπουμε ότι είναι αρκετά σημαντικός τομέας κυρίως για παραμεθόριες περιοχές, γειτονικές μεταξύ τους περιοχές, με πολλά ωφέλη. Θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα το τι συμβαίνει, γι' αυτό ε, παραγγείλαμε μελέτες που εκδόθηκαν το Μάρτιο, και εκεί παρέχονται template, παρέχονται κουτίκια εργαλείων και παραδείγματα καλή καλής συνεργασίας. Τι η μελέτη στις 4 Δεκεμβρίου θα προβληθεί και θα παρουσιαστεί και σε μια σχετική διάσκεψη για την υγειονομική περίθαλψη των διασυνοριακών περιοχών που διοργανώνουν από κοινού η DG Sante και Ρίτζιο. Και τα σημαντικά εργαλεία συνεργασίας μας που προβλέπονται και από αυτήν την οδηγία είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Share, care and cure, δηλαδή μοιραζόμαστε, ε, παρέχουμε φροντίδα και θεραπεύουμε. Ένα σημαντικό δίκτυο που συμμετέχουν 500 γιατροί, ασθενείς, ε, διευθυντές νοσοκομείων, εκπρόσωποι ενός ασθενών. Ήρθαν στις την περασμένη εβδομάδα μάλιστα. Συζητήσαμε το πώς προχωράνε τα πράγματα και τι πρέπει να γίνει. Αναφέραμε και το δίκτυο με τις 950 τεχνολογικά εξοπλισμένες μονάδες οικονομικής περίθαλψης, εκατοντάδες νοσοκομεία και ιατρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολλές οι υπηρεσίες ιατρικές που συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο και σε αυτή τη φάση δεν σκοπεύουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των δικτύων, διότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τα ήδη υπάρχοντα. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο ρήμανσης τώρα και θα πετύχουμε, πιστεύουμε, τους στόχους μας. Για την ηλεκτρονική υγεία, την υγεία ψηφιακά, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιχειρήσει την ε, ηλεκτρονική μετατροπή πολλών συστημάτων βάσει και τη απόφαση που δημοσιεύτηκε το 2018. Εργαζόμαστε για το ηλεκτρονικό δίκτυο υγείας που απαιτείται και από αυτή την οδηγία. Και προσπαθούμε και εδώ μαζί με τα κράτη-μέλη να βρούμε το κατάλληλο τρόπο διαχείρισης. Και πώς θα έχουμε την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Σημαντικό είναι να πούμε ότι 22 κράτη-μέλη συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα διευκόλυνσης της διασύνδεσης της Ευρώπης και ελπίζουμε ότι του χρόνου θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή συνταγογραφήσεων μεταξύ 100 μελών έστω και ανεπισήμως, ατύπως. Για να ολοκληρώσω, είναι πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς μας αυτό. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζουμε να επιδιώκουμε οι πληροφορίε να φτάνουν στα αυτιά των πολιτών, αλλά όπως είπαν και διάφοροι ομιλητέ. η γνώση ταξιδεύει καλύτερα όταν όντω ωφελούνται από όλα αυτά τα εργαλεία μα οι ίδιοι ασθενεί και οι εργαζόμενοι στον τομέα τη υγεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπέλετ. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και συνοψίζοντας να πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ένα μεγάλο εγχείρημα αυτό, μια πλατφόρμα με κοινού στόχους, όπως εκφράστηκαν και εδώ, η έλλειψη ενημέρωσης. Είναι δική μας αρμοδιότητα και καθήκον να αυξήσουμε το επίπεδο γνώσης. Το πώς λειτουργούν τα εθνικά σημεία επαφή και να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχουν. Το είπε και η κυρία Ρης, από το 10% πρέπει να πάμε στο 90%. 90 θέλουμε να φτάσουμε. Όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζουν και τα δικαιώματά τους και ότι υπάρχει μια ενιαία θηρίδα, απευθυντική. Και για την επιστροφή των εξόδων και για τις αποζημιώσεις, για τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις και το καθεξής. Η σημασία της ηλεκτρονικής υγείας το είπε και η κυρία Ρή, είπε για το ψήφισμα που εγκρίναμε και συνδέεται άμεσα με αυτό που τώρα μας αποσχολεί. Δεν μπορούμε να μιλάμε για διασυνοριακή υγεία εάν δεν λάβουμε υπόψη μα και την ηλεκτρονική υγεία που είναι μια εξέλιξη για να μην πω επανάσταση. Ο κύριος λέει, είπε ότι οι φιλοδοξίες μας θα πρέπει να είναι ε, φιλοδοξίες κυκλοφορίας, έντονης κινητικότητας των ασθενών. Πρέπει πρώτα όμως να φροντίσουμε την κυκλοφορία της γνώσης και των πληροφοριών. Γι' αυτό και η ηλεκτρονική υγεία, οι συνταγογραφήσεις, πρέπει όλα αυτά να διευκολυνθούν και να προωθηθούν. Η σημασία των παραμεθόριων περιοχών είναι σημαντικές, το είπε ο κ. Πέτρελε, και ο κύριος Ρίσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις, παραδείγματα και καλή συνεργασία μεταξύ γειτονικών περιοχών, πιο συγκεκριμένα όταν μιλάμε για τις ηλεκτρονικές συνταγές. Πιο σημαντικές είναι ακριβώς για αυτές τις περιοχές που είναι παραμεθόριες και γειτονικές. Τα σχολεία σα, είπε ο κ. Βόλκε, την έλλειψη πληροφοριών και του σαφεί κανόνε για την επιστροφή των εξόδων. Όσο υπάρχουν ε, όσο υπάρχει σύγχυση και έλλειψη γνώση για το αν ε, επιστρέφονται τα έξοδα ή όχι, ασθενεί δεν θα πάνε ούτε στη δίπλα γειτονιά. Οπότε πρέπει να είναι σαφέ το τι ισχύει οικονομικώ για τη διασυνοριακή υγεία. Και η κυρία Σράγερ είπε ότι το μέγεθος του προβλήματος αυτού είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε εντοπίσει για την ώρα. Είναι θέμα διαθεσιμότητας φαρμάκων, διασυνοριακά. πρέπει και αυτό να μας απασχολήσει και να το κοιτάξουμε. Έχοντας φυσικά υπόψη ότι οδεύουμε προς τις ευρωεκλογές. Πάνω απ' όλα η υγεία και η υγειονομική περίθαλψη απασχολεί του πολίτες. Είναι πρόβλημα, είναι θέμα που του νοιάζει. Οπότε πρέπει να ε, ξεκαθαρίσουμε κι εμείς ότι υπάρχει προσδεθέμενη αξία χάρη στην ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ γειτονικών περιοχών ε, που είναι και παραμεθόριες. Ε, share, care and cure. Μοιραζόμαστε, φροντίζουμε και θεραπεύουμε. Το είπαν και η κυρία Ρης και ο κύριο Ρης τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αυτά είναι τα πιο σημαντικά και καλύπτουν και τι ανησυχίε του κυρίου Πέτρελε, την κυκλοφορία των ασθενών. Κυκλοφορία των ασθενών και κυκλοφορία των γνώσεων. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχο μα, οπότε προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία με του Κιώδη. Μόλι ε, εκπνεύσει και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, θα φροντίσουμε να συναντηθούμε για να βρούμε και συμβαστικέ. Θα συνεδριάσουμε σύντομα. Ευχαριστούμε. Να σας θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 4 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΝΒΙ τον Ιανουάριο, 21 και 22 του μήνα. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι τροποποιητικός κανονισμός Τη κοινή Γεωργική Πολιτική ε, και συντάκτη τη Νομοδότηση είναι ο κύριο Ντόρφμαν, τον οποίο αντικαθιστά σήμερα η κυρία Κατίνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας μεταφέρω τη συγνώμη του συναδέλφου Ντόρφμαν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι εδώ και ζητά να τον, να τον συγχωρείτε μου ζητά σύντομα να παρουσιάσω τη σχέδιο γνωμ... εκθεσής του, γνωμοδότησής του. Πρόκειται για ένα κείμενο που απευθύνεται στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου για την πρόταση κανονισμού που αλλάζει την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών. Στη φάση αυτή, το κείμενο που θα σας διαβάσω για λογαριασμό του συναδέλφου Ντόρφμαν επικεντρώνεται στις αρμοδιότητες της δικής μας ε, Επιτροπής του Περιβάλλοντος. Τρία είναι τα σημεία που πρέπει να σας διαβάσω. Πρώτον, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει τη δυνατότητα της ε, συνέχισης της καλλιέργειας της Βήτης Λαμπρούσκα και προβλέπει και την δυνατότητα καλλιέργειας άλλων ε, υβριδικών ποικιλιών. Για τις νέες ποικιλίε αμπέλου, ο εισηγητής ε, δέχεται τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα υβριδικά. Αλλά ενώ η, ή μάλλον η έκθεση του, του συναδέλφου Ντόρφμαν περιορίζει την καλλιέργεια των παλιών ποικιλιών, της Β. Λαμπρούσκα συγκεκριμένα, δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να την εγκρίνουν, αλλά μόνο για ιστορικούς λόγους. Εάν δεν υπάρξει αύξηση και αν δεν υπάρξει μέλλον και αύξηση στι καλλιεργούμενε εκτάσει. Οπότε εντάξει η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι νέε ποικιλίε, αλλά σε ό,τι αφορά τι παλιέ, να αποφασίζουν τα κράτη-μέλη αν θα δώσουν έγκριση ή όχι, αλλά η έγκριση να δίνεται μόνο για ιστορικούς λόγους, για λόγους παράδοσης. Και ε, στο μέγεθος και στην έκταση που ήδη καλλιεργείται το είδος αυτό. Έπειτα, σε ό,τι αφορά την ετικετοθεσία, την επισήμανση, ο συνάδελφος Ντόρφμαν, συμφωνώντας με τον κανονισμό 1669 του 2011, ζητά από τον παραγωγικό τομέα να σέβεται την ενεργειακή αξία από την παραγωγή και την καλλιέργεια αμπέλου. Ε, στο τρίτο σημείο, η συγκεκριτή στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, τα, για τους ίνους χωρίς ε, περιεκτικότητα σε αλκοόλ ή μερικώς ε, χωρίς αλκοόλ. Αυτά δεν είναι κρασιά τα οποία προστατεύονται από γεωγραφική ένδειξη. Σύμφωνα με τον εισηγητή, είναι σωστό να επιτρέψουμε την αφαίρεση του αλκοόλ από, τα, από τους ίνους εκεί όπου επιτρέπεται η αντίθετη διαδικασία, δηλαδή εφόσον κάποιοι αυξάνουν την περιεκτικότητα σε αλκοόλ των κρασιών. Όμως θεωρεί ότι τα κρασιά αυτά μπορεί να ανοίξουν νέες αγορές για, τις, ε, για τους ευρωπαϊκούς ίνους. Αυτά είναι τα κεντρικά σημεία. Και για να ολοκληρώσω, τα τρία αυτά σημεία του σχεδίου γνωμοδότησης εννοείται ότι ο συνάδελφος Ντόρφμαν είναι στη διάθεσή σας για να τα συζητήσει περαιτέρω μαζί σας και να δείτε και τις λεπτομέρειες μαζί του. Σας ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας στη συζήτηση. Ευχαριστούμε. Τώρα οι σκιώδεις, οι αντικαταστάτες τους. Ο κύριος Βόλκεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο κύριος Καπούτο είναι ο σκιώδη εισηγητής δεν μπορεί να είναι παρόν και γι' αυτό θα διαβάσω μία δήλωση εκ μέρου του. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι ιδιαίτερα εκτενή και έχει να κάνει με την κοινή οργάνωση αγοράς για γεωγραφικά προϊόντα και έχει να κάνει επίσης με τις γεωγραφικές ενδείξεις ε, των αρωματισμένων αμπελοϊνικών προϊόντων και επίση έχει να κάνει με τι αξόχω ε, απόκεντρε περιοχέ και τα μικρά νησιά. Ο κύριος Καπούτο θέλει να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις πτυχέ που αφορούν την Επιτροπή ΕΝΒΗ. Καταρχά, ε, όσον αφορά ε, την επισήμανση με τα θρεπτικά στοιχεία, οι πληροφορίε ε, σχετικά με τις θερμίδες και τα συστατικά του ίνου πρέπει να γίνεται, διότι οι καταναλωτέ ε, έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πόσε θερμίδε καταναλώνουν όταν πίνουν ένα ποτήρι κρασί. Και γι' αυτό ε, χαίρεται πολύ με τα βήματα που έχουν γίνει από τον τομέα του ίνου τους τελευταίους μήνες. Οι ε, ινοπαραγωγοί είναι διατεθειμένοι να αναφέρουν τον αριθμό θερμίδων στο, στις φιάλες και ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τη την επιθυμία αυτή, τη βούληση αυτή. Ε, επίσης, ο κύριος Καπούτο πιστεύει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, τις οικονομικές συνέπειε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι άλλωστε η σπονδυλική στήλη του αμπελοϊνικού τομέα στην Ευρώπη θα πρέπει οι πληροφορίες να μπορούν να δίδονται και με ψηφιακή μορφή. Όσον αφορά τα υβρίδια και ε, τη, τα κρασιά με γεωγραφική ένδειξη, ο κύριος ε, Καπούτο συμφωνεί, αλλά δεν συμφωνεί να γίνεται χρήση των ε, έξι απαγορευμένων ποικιλιών στα κράτη-μέλη, διότι αυτές οι ποικιλίε Ε, δεν είναι ενδιαφέρουσες ε, από οργανοληπτικής άποψης. Επιπλέον, έχουν απαγορευτεί από τη δεκαετία του 1930 λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε μεθανόλη, κάτι που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους καταναλωτές. Ο κύριος Καπούτο πιστεύει ότι, οι ότι απαιτούνται επιστημονικές μελέτες ε, όσον αφορά την ε, χρήση της ποικιλία ε, βήτης λαμπρούσκα. Επίσης δεν συμφωνεί με την τροποποίηση του ορισμού σχετικά με τις προστατευμένες γεωγραφικές ενδείξεις. Προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τονιστεί η ανθρώπινη πτυχή, αλλά αυτό δεν συνάδει με τον ΠΟΕ θα πρέπει να υιοθετήσουμε τον ορισμό του ΠΟΕ. Και τέλος, σε αντίθεση με τον εισηγητή κύριο Ντόρφμαν, ο κύριος Καπούτο πιστεύει ότι ε, οι ίνοι χωρίς αλκοόλ δεν μπορούν να, να υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς με τα κανονικά κρασιά. Αυτό άλλωστε έχει να κάνει με το παράρτημα 7 τμήμα 2 της κοινή οργάνωσης αγοράς. Ε, τα εθνικά προγράμματα στήριξης προορίζονται μόνο για γεωργικά προϊόντα και όχι για βιομηχανικά. Ο κύριος Καπούτο θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ανταποκριθούμε στο αίτημα των καταναλωτών για διαφάνεια και να μην ε, δημιουργούμε ε, παρεξηγήσεις. Ε, τέλος, ε, θέλει να καλέσει τους ε, ε να ασχοληθούν με το θέμα της απόσταξης και των καταλήπων. Ο κύριος Καπούτο θέλει τα σχετικά πλεονεκτήματα να διαβρινθούν και στην κομποστοποίηση, κάτι που μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Για παράδειγμα, η ενέργεια που προέρχεται από την μεθανοποίηση να ε, εισάγεται στα εθνικά δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Γιατεμάκη, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένη με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αναδιοργάνωση ε, του κανονισμού. Αυτό είναι κατανοητό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που ζητάει περισσότερες πληροφορίες ε, στην επισήμανση των ίνων. Όπως και οι προλαλήσαντες, θεωρώ και εγώ ότι είναι σημαντικό οι καταναλωτές να έχουν περισσότερες πληροφορίες ε, σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση κατά την παραγωγή. Το, είναι τώρα αυτός ο κατάλληλος κανονισμός ε, για κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτα σαφές. Όσον αφορά την επισήμανση, καταλαβαίνω ε, ότι η γεωγραφική ένδειξη είναι ευαίσθητο θέμα, ωστόσο πρέπει να προσαρμόσουμε τη γεωργία μας στην ε, αλλαγή του κλίματος, εισάγοντας νέες ποικιλίε ίνου. Παρότι δεν είναι εδώ ο εισηγητής, ε, θα ήθελα τέλος ε, να ακούσω καλύτερη αιτιολόγηση σχετικά με το γιατί διευρύνει τον κανονισμό ως, το, ως προς τις ποικιλίε, διότι δεν έχω ακόμη καταλάβει περί τίνο πρόκειται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω εδώ έχουμε να κάνουμε ε, με έναν όχι και τόσο συναρπαστικό τομέα της ε, μεταρρύθμισης του, της κοινή γεωργικής πολιτικής. Έχει να κάνει με την κοινή οργάνωση αγοράς ε, και γενικά είμαι σύμφωνος με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τις τροπολογίες του κυρίου Ντόρφμαν, τίθεται το ερώτημα γιατί να πρέπει να περιοριστούμε στις παλιές ποικιλίε. Δεν ξέρω αν είναι καλή η πρόταση το, όπως ε, έχει υποθεί και στην Επιτροπή Γεωργίας ε, το να ε, έχουμε η ίδια μεταχείριση και στα κρασιά όπου έχει, αφαιρεθεί, όπου έχει αφαιρεθεί μέρος της αλκοόλης. θα πρέπει να φροντίσουμε να, να μην χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια στην, στον κανονισμό αυτών. Εδώ στην πρόταση μιλάμε για τον ίνο που είναι πολύ ενδιαφέρον και επίμαχο θέμα σε κάποιες περιφέρειες. Αλλά ε, σκεφτείτε και τον τομέα του γάλακτος. Θέλουμε να ενισχύσουμε Ε, τον τομέα αυτών. Ε, θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τι ε, προϋποθέσεις μπορούμε να προσφέρουμε στον τομέα των γαλακτοκομικών. Θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να πάρει το λόγο πάνω στο θέμα αυτό. Εάν όχι, να δώσω το λόγο στον κύριο Σέρα εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, συμβολή του στην ε, αναθεώρηση των ε, κανόνων αυτών, στον τροποποιητικό κανονισμό δηλαδή, που τροποποιεί τον διάφορους κανονισμούς. Βλέπω ότι ο εισηγητή είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, δοθεί τέλος ε, σε απαγόρευση κάποιων ποικιλίων και ιδιαίτερα όσον αφορά την ποικιλία βιτης Λαμπρούσκα. Έχει λιγότερο φιλόδοξη προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ συμφωνεί απολύτω με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τι απογορευμένε ποικιλίε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η παραδοσιακή πολιτική όσον αφορά την σε βινήφερα δεν αιτιολογείται πια από τις σημερινές συνθήκες. Σήμερα έχουμε επιστημονικά τεκμήρια που δείχνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και γι' αυτό δεν αιτιολογείται και η σχετική απαγόρευση. Θα είναι χρήσιμο να εισάγουμε πιο ανθεκτικές ποικιλίε με στόχο τη μείωση και των φυτοπαφαρμάκων μέχρι 80% σε σχέση με την ποικιλία β της βινήφερα. Ξέρω ότι ο εισηγητής, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύει ότι ε, είναι από τους οποίους έχει αφαιρεθεί μέρος της αλκοόλης ή η αλκοόλη. Ε, δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι έτσι μπορούμε να προσαρμοστούμε καλύτερα στις αγορές ίνου του παρόντος και του μέλλοντος. Γι' αυτό θα είναι χρήσιμο να μπορούμε να προσφέρουμε στους συνοπαραγωγούς όλα τα απαραίτητα μέσα για να παραμένουν ανταγωνιστικοί, προστατεύοντας παράλληλα και τον καταναλωτή με σωστή επισήμανση των ε, νέων αυτών κατηγοριών προϊόντων. Ξέρω ότι ο η στην πρότασή του έχει συμπεριλάβει το πολύ ε, ευαίσθητο θέμα της επισήμανσης ε, και του κατάλογου συστατικών των ίνων, ενώ, όπως όλοι γνωρίζουν, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουνίου του 2018 δεν περιλαμβάνει σχετική πρόταση. Αυτό όμως ε, δεν οφείλεται στο ότι δεν πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά στοιχεία αυτά. Αντιθέτως, κατά την υιοθέτηση της πρότασης ε, είχαμε μια παράλληλη διαδικασία που ξεκίνησε με την έκθεση της ε, Αρμόδιας Επιτροπής για την επισήμανση των ε, ίνων ε, και άλλων ποτών που κάλυπτε τον τομέα αυτό στο σύνολό του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει ακόμη την έκθεση αυτή και βλέπουμε ότι ο αμπελοϊνικός τομέας θέλει τομεακή προσέγγιση, δηλαδή να έχουμε μια σειρά κανόνων που να ισχύει για το κρασί. Επικροτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θάρρος της, ε, του αμπελοϊνικού τομέα που ζητάει περισσότερη διαφάνεια στην επισήμανση. Γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει με ενδιαφέρον κάθε τομεακή πρόταση που θα μπορούσε να προκύψει από το Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Ταυτόχρονα, άσχετα από το νομικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί, είναι σημαντικό να πετύχουμε το διτό μας στόχο, δηλαδή να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή από τη και από την άλλη να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Καρδίνη, αν έχει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ. Προφανώς θα φροντίσω να αναφέρω όσα συζητήθηκαν σήμερα εδώ μεταξύ μας, τον συνάδελφο Ντόρφμαν και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το θέμα. Εισηγητής, παρόλα αυτά, συνεχίζει να είναι εκείνος. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 29 Δεκεμβρίου στις 12 και θα ψηφίσουμε στις 29 Ιανουαρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα πολύ χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Χαντσποφλέρ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την ειδική έκθεση του IPCC για την παγκόσμια θέρμανση 1,5 βαθμού Κελσίου. Είναι πρόεδρο τη ομάδα εργασία 2 του IPCC από το 2015. Η ομάδα αυτή εργασία επικεντρώνεται στι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή εντοπίζει πόσο ευάλωτα είναι τα κοινωνικά και φυσικά συστήματα στην κλιματική αλλαγή και τι επιπτώσεις υπάρχουν. Εξετάζει με ποιο τρόπο οι άνθρωποι μπορούν να προσαρμοστούν στην θέρμανση του πλανήτη. Ο καθηγητής Πόλνερ έχει μεγάλη εμπειρία στις δραστηριότητες του IPCC ήταν ε, υπεύθυνο για την πέμπτη έκθεση που ολοκληρώθηκε το 2014 εν ώψη των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία των Παρισίων. Με τη Συμφωνία των Παρισίων, λοιπόν, που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015, 195 χώρες συμφώνησαν να περιορίσουν την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους δύο βαθμούς ε, Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να περιοριστεί αυτή η αύξηση σε 1,5 βαθμό Κελσίου. Μέρος της συμφωνίας οι κυβερνήσεις κάλεσαν ε, το IPCC να ετοιμάσει μια ειδική έκθεση το 2018 για τις επιπτώσεις της ε, θέρμασης του πλανήτη 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και τη σχέση με την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου. Ολοκληρώθηκε εκθέ τον Οκτώβριο του 2018 και τώρα έχει ξεκινήσει διάλογος, ο διάλογος του Ταλανόα, όπως ονομάζεται. Θα μπορέσουμε λοιπόν να συζητήσουμε εδώ μεταξύ μας. Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας, κύριε καθηγητά, και σας δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι εδώ και να σας μιλήσω για την ειδική μας έκθεση όσον αφορά τη θέρμανση του πλανήτη κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Θα σας μιλήσω βέβαια από το πρίσμα των επιπτώσεων, τα ωφέλη δηλαδή αν η θέρμανση αυτή γίνει 1,5 βαθμό αντί για 2 βαθμούς. Γιατί ακριβώς οι επιπτώσεις είναι που καθοδηγούν τις φιλοδοξίες μας προκειμένου να υπάρξει η άμβληση του φαινομένου και προσαρμογή. Η έκθεση αυτή λοιπόν προσθέτει την άλλη μας έκθεση που έχει γίνει για τους δύο βαθμούς Κελσίου και γίνεται σύγκριση με τον 1,5 βαθμό. Το ερώτημα είναι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά τις επιπτώσεις. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαφορά στη συμπεριφορά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί έτσι η Συμφωνία των Παρισίων έτσι γίνεται περισσότερο κατανοητή. Οι επιπτώσεις λοιπόν με την αύξηση κατά 1,5 βαθμό θα οδηγήσει σε λιγότερα κρέα καιρικά φαινόμενα εκεί που οι άνθρωποι ε, ζουν και θα υπάρχει λιγότερο υπερβολική ζέστη, καύσονες και λιγότερες βροχοπτώσεις, υπερβολικές βροχοπτώσεις. Επίσης το 2100 το επίπεδο της ε, θάλασσας θα έχει ε, αυξηθεί κατά 10 εκατοστά λιγότερο. Κάτι το οποίο βεβαίως και κάνει διαφορά και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αύξηση αυτή του επίπεδου της θάλασσας μπορεί να συνεχιστεί και για αιώνες μετά το 2100. Αυτό είναι γνωστό στην επιστημονική κοινότητα ότι κάθε μήνα αυξάνει το επίπεδο της θάλασσας. Επίσης, ε, κατά 10 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι θα εκτίθεται στον κίνδυνο αυτό της αύξησης του επίπεδου της ε, θάλασσας μέχρι το 2018 και θα κινδυνεύουν λιγότερο και τα παράκτια οικοσυστήματα. Το ερώτημα βέβαια είναι πού θέλουμε να πάμε εφόσον μιλάμε για 1,5 βαθμό αντί για 2 βαθμούς χαμηλότερη επίπτωση στη βιοπικιλότητα και στα διάφορα είδη. Επίσης, πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο, μικρότερη μείωση της ε, σοδιάς του ρυζιού, ε, σιτηρών. Ο συνολικός ο πληθυσμός επίσης που θα κινδυνεύει να μην έχει αρκετό νερό θα είναι κατά 50% λιγότερο με 1,5 βαθμό αντί με 2 και άρα θα υπάρχει και λιγότερο πρόβλημα ίδρευσης για τα οικοσυστήματα. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στο χερσαίο χώρο, αλλά εδώ έχω βάλει και μία διαφάνεια για τις θάλασσες και τι βλέπουμε εδώ συγκρίνοντας τους δύο με τέσσερις, πέρα δηλαδή από αυτά που λέει η έκθεση. Αυτό που βλέπετε, η γκρίζα ζώνη δηλαδή, δείχνει ότι θα υπάρξει μεγάλη απώλεια βιοπικιλότητας. Κάτι το οποίο έχει να κάνει με ευαίσθητα συστήματα, κοραλιογενείς περιοχές κτλ. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για ορισμένους χώρους. Βλέπετε ότι και στο Βόρειο Πόλο επίσης. Και η θέρμανση και η ταχύτητα με την οποία αυτή λαμβάνει η χώρα κάνει τη διαφορά. Αν συνεχίσουμε τη σύγκρισή μας, 1,5 βαθμοί Κελσίου σε σχέση με τους δύο, ε, με τον 1,5 βαθμό θα έχουμε λιγότερο κίνδυνο για την αλία. Γιατί πολλές χώρες εξαρτώνται από την μικρή κλίμακα σαλία. 700 εκατομμύρια λιγότεροι θα κινδυνεύουν ε, από προβλήματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και άρα και με μεγάλη φτώχεια μέχρι το 2050. Άρα πρόκειται εδώ πέρα και για κοινωνικά φαινόμενα που παίζουν ρόλο ανάλογα με το αν θα έχουμε 1,5 ή 2 βαθμούς αύξηση. Θα επεκταθώ περισσότερο σε αυτό αργότερα. Πάντως με 1,5 βαθμό αντί για 2 Ήδη οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την Αρκτική, για τις άνυδρες ε, ζώνες, για μικρά νησιά αναπτυσσόμενων χωρών. Οι άνθρωποι εκεί είναι πάρα πολύ ευάλωτοι. Με 1,5 βαθμό αντί για 2, επίσης υπάρχουν λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία, για να έχουμε αρκετά τρόφιμα, ε, νερό, πόσιμο και θα υπάρχει περισσότερη ασφάλεια για τον άνθρωπο και οικονομική ανάπτυξη. Ε, βέβαια υπάρχουν ε, διάφορα στοιχεία προσαρμογής που μπορούμε να υιοθετήσουμε για να περιορίσουμε τις κλιματικούς κινδύνους. Αλλά βέβαια αυτή η προσαρμογή χρειάζεται σε λιγότερο βαθμό εφόσον η αύξηση είναι 1,5 βαθμό αντί για 2. Εδώ πέρα βλέπουμε τις επιπτώσεις σε σχέση με τον κίνδυνο και έχουμε επιλέξει εδώ πέρα διάφορα χρώματα για να αναλύσουμε και να αξιολογήσουμε αυτούς τους κινδύνους. Και κάτω δεξιά βλέπετε τον ε, κώδικα αυτό. Έχουμε τον κίνδυνο που δεν εντοπίζεται μέχρι μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο. Για την κάθε κατηγορία κινδύνου υπάρχει μια εξήγηση που περιγράφει το τι μπορεί να συμβεί κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι λόγια ανησυχία που εξηγήσαμε και σε προηγούμενες εκθέσεις μας, μόνο που εδώ υπάρχουν διαφορετικά όρια εξαιτίας των νέων στοιχείων που διαθέτουμε για τις επιπτώσεις. Έχουμε λοιπόν συστήματα τα οποία απειλούνται πάρα πολύ, όπως είναι οι καλλιεργενείς ε, περιοχές ή η Αρκτική. Η βιοπικιλότητα κινδυνεύει πολύ. Εδώ βλέπετε τη σύγκριση ανάμεσα στον 1,5 βαθμό και τους 2 βαθμούς και σε μερικές περιπτώσεις είμαστε ήδη σε υψηλό κίνδυνο και με τον 1,5 βαθμό, αλλά βέβαια ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος με τους 2 βαθμούς. Κυρίως για μοναδικά συστήματα, αλλά όχι μόνο. Έπειτα έχουμε το θέμα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυξάνονται οι ζημιές, οι απώλειες, εφόσον έχουμε ε, ακραία καιρικά φαινόμενα, θύελες, πλημμύρες κλπ. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα έχουμε όλο και περισσότερο. Και το τέλος είναι κάποια μεμονωμένα γεγονότα, τα οποία έχουν να κάνουν με την ε, κατάρρευση των πάγων στο Βόρειο Πόλο και την αύξηση του επίπεδου της θάλασσας. Εδώ υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα. Μπορούμε όμως να πούμε ότι ο κίνδυνος ε, αυξάνει όσο έχουμε μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη. Ένα άλλο παράδειγμα που έχουμε είναι εδώ από την Αρκτική. Εδώ συγκρίνουμε πάλι τον 1,5 βαθμό με τους 2 αύξηση. Με 1,5 θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ε, κάποιους πάγους στην Αρκτική, ενώ εφόσον η αύξηση της θερμοκρασίας είναι δύο βαθμοί, εδώ θα είναι πολύ πιο δύσκολο, πολύ λιγότεροι πάγοι θα διατηρηθούν. Και βέβαια έχει να κάνει και με το οικοσύστημα. Βλέπετε εδώ πέρα ένα ζωικό είδος, αλλά η θέρμανση της Αρκτικής έχει επιπτώσεις στο κλίμα γενικότερα με αποτέλεσμα ακραία καιρικά φαινόμενα και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Εξαιτία τη διαφορά στη θερμοκρασία δηλαδή ανάμεσα στην Αρκτική και άλλα μήκη και πλάτη. Αν πάμε πιο πέρα για την αξιολόγηση κινδύνου και θέλουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πρέπει πάνω απ' όλα να δούμε τι γίνεται στις κορυλογενείς ε, θαλάσσιες περιοχές που μειώνονται εξαιτία της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό βέβαια με άλλα φαινόμενα. Είμαστε σε υψηλά επίπεδα κινδύνου έως πολύ υψηλά επίπεδα κινδύνου. Δηλαδή χάνουμε μεγάλες επιφάνειες κοραλιογενείς. 70 με 90% θα χαθούν ακόμα και με 1,5 βαθμό Κελσίου αύξηση. Θα χάσουμε επίσης και την εξυπηρέτησή τους σε, στον άνθρωπο, στην αλία κλπ. Μπορεί να μην εξαφανιστούν τελείως, αλλά το ωφέλη για τον άνθρωπο θα μειωθούν πολύ. Μετά βλέπουμε την Αρκτική, εδώ στην τελευταία διαφάνεια πάλι βλέπουμε την αλλαγή που πηγαίνουμε από υψηλά σε πολύ ψηλά επίπεδα κινδύνου σε διάφορες περιπτώσεις, στις πλημμύρες, στις ακτές. Και κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρέπει να μιλήσουμε και για τη θνησιμότητα εξαιτίας των υπερβολικά ψηλόθερμοκρασών, καυσών δηλαδή που έχουμε σε διάφορες χώρες και σε διάφορες περιοχές. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για τον θάνατο των ανθρώπων που έτσι κι αλλιώς πεθαίνουν περισσότερο και ο κίνδυνος θα αυξηθεί από μέτριο σε υψηλό με δύο βαθμούς θέρμανση αντί αλλά έχει να κάνει και με το ζωικό βασίλειο, που επίσης επηρεάζεται από τους καύσονες γιατί η ζωή τους εξαρτάται, όπως και των ανθρώπων, από την ρύθμιση της θερμοκρασίας. Συνεπώς, ήδη έχουμε ζημιά με τον 1,5 βαθμό, αλλά λιγότερη από ό,τι θα είχαμε με τους 2 βαθμούς. Τώρα, τι γίνεται με τις κορελογενείς περιοχές και τι έχουμε διαπιστώσει στις τελευταίες μας αξιολογήσεις. Εδώ βλέπουμε τη διαφορά. Στα αριστερά βλέπετε μια ε, κορολογενή περιοχή που βρίσκεται σε πλήρη υγεία. Στη μέση βλέπουμε πώς αλλάζει η κατάσταση εξαιτία της θέρμανσης των υδάτων. Χάνονται κάποια είδη. Αν λοιπόν η υπερθέρμανση αυτή είναι περιορισμένη στο χρόνο, τότε ανακάμπτει το είδος. Αν όμως η υπερθέρμανση αυτή κρατήσει πολύ, τότε πεθαίνουν αυτά τα είδη και ο βυθός γίνεται μια έρημος που γεμίζει από φύκια και δεν μπορεί να ανακάμψει. Αυτά συμβαίνουν ήδη και πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την καταστροφή αυτή όσο μπορούμε περισσότερο. Αν δείτε την εικόνα από το διάστημα, ήδη το 2016 ο κίνδυνος είχε ήδη αυξηθεί και στην Αυστραλία, για παράδειγμα, χάθηκε άλλο 90% του περιθωρίου που υπήρχε με τον 1,5 βαθμό. Συνεπώς πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και πώς η έκθεση ήδη υπογραμμίζει τη διέξοδο που έχουμε και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Τα πιο φιλοδόξα σενάρια τα βλέπετε πάνω αριστερά και τα πεσιόδοξα κάτω δεξιά. Βλέπετε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των διαφόρων ε, υποθέσεων αυτών στα πάνω διαγράμματα δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου κίτρινα. Ε, το κίτρινο έχει να κάνει με τη διαδικασία που ονομάζουμε DEX, τη χρήση της βιοενέργειας που συνδυάζεται με την αποθήκευση και τη διατήρηση του άνθρακα για να αντιμετωπίσουμε την ύπαρξη υπερβολικά πολύ διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Εδώ ε, αυτό επηρεάζει τη βιοπικιλότητα, την επιστημιστική ασφάλεια για την ανθρωπότητα και για τα ζωικά είδη, διότι υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό με την, ε, μεταξύ γεωργία, παραγωγή τροφίμων για, τα, για του ανθρώπου και τη φύση. Όσο λιγότερο τηρούμε τι υποχρεώσει εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, τόσο ε, περισσότερο δεν εφαρμόζουμε τεχνολογίε όπω η DEX που τη χρειαζόμαστε. Τα τροπικά δάση θα ήταν αρκετά για αν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι ώστε στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε την υπερθέρμανση στο 1,5. Αυτή λοιπόν η διαφορά με τον DEX είναι καθοριστική. Όσο περισσότερο περιμένουμε για να αναλάβουμε φιλόδοξη δράση, τόσο περισσότερο θα επαφιόμαστε σε αυτήν την τεχνολογία φιλόδοξη μείωση των ε, εκπομπών ε, ελαχιστοποιεί την ανάγκη για την ε, απαλλαγή από τον άνθρακα και τα διοξίδια του και έχει πολλά ωφέλη για την ανθρωπινή υγεία, για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και την αποθήκευση του διοξιδίου με την διοπικιλότητα να διατηρείται και λιγότερο ανταγωνισμό για τη γη ε, και τη χρήση της για την παραγωγή τροφίμων ή για την κατοικία της ανθρωπότητας. Τελευταίο, θα πρέπει να σκεφτούμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ε, κλήσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη από τον ΟΗΕ ότι μπορούμε να έχουμε ένα συνολικό συμπέρασμα από την έκθεση για το 1,5 για τον 1,5 βαθμό. 1,5 ε, βαθμός θα πει ότι μπορεί και να πετύχουμε τους στόχους της χιλιετίας, αν καταφέρουμε να το κρατήσουμε εκεί. Και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν πολλοί τομείς που μπορούν να συνεργαστούν ε, σε αυτό, όπως η παροχή ενέργειας, η ζήτηση ενέργειας, η χρήση της γης, τα γαλαζοπά χρώματα, λένε πώς η πραγματική δράση αναχέτησης μπορεί να συνδυαστεί και να ωφελήσει ανάπτυξη. τον αντίστοιχο στόχο βιώσιμη ανάπτυξη. Πάνε σε ζεύγη. Βλέπετε ότι συνολικά υπάρχουν αμοιβαία ωφέλη για, όλες, για όλους τους τομείς, εάν παραμείνουμε στο 1,5 βαθμό και δεν φτάσουμε στους 2. Και είναι πολύ λίγα τα μειονεκτήματα της χρήσης αυτών των τεχνολογιών. Ωστόσο, βλέπετε και θα το έχετε ζήσει κιόλα, ε, θα το έχετε καταλάβει ήδη από την παρουσίαση, ότι 1,5 βαθμός ε, δεν είναι και καμένας παράδεισος και καμιά ιδανική λύση. Είναι συμβαστική λύση μεταξύ του ότι είναι εφικτό και τι είναι ρεαλιστικό. Υπάρχουν όμως και κάποια... Ε, ε κόλπα, περίεργα σημεία που πρέπει να τα επιλύσουμε για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Δηλαδή ε, το κατά πόσον οι μόνιμοι πάγοι και οι εκτάσεις τους προστατεύονται για να μην αυξηθεί κι άλλο η στάθμη της θάλασσας. Θα παραμείνουν ε, ως έχουν. Η έρευνα θα μας τα πει αυτά. Προς στιγμήν φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημείο όπου θα αλλάξουν δραστικά τα πράγματα μεταξύ του 1,5 βαθμού και των 2 βαθμών. Αλλά αν η στάθμη της θάλασσας αυξη, ε, ξεφύγει από αυτό το όριο το συγκεκριμένο, μπορεί να ε, αυξηθεί πολύ η στάθμη της θάλασσας, μέτρα ολόκληρα και όχι απλώς μερικά εκατοστά. Μπορεί δηλαδή να ζούμε σε έναν πολύ επικινδυνότερο κόσμο, ακόμη και αν επιλέξουμε τον 1,5 βαθμό ως στόχο. Αυτές οι τιμές ε, είναι πολύ κοντινές στις, ε, στα ευρήματά μας για την προϊστορία, για το τι συνέβαινε πριν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, όταν η θερμοκρασία του πλανήτη ήταν περίπου παρόμοια με τη σημερινή και η στάθμη της θάλασσας ήταν 5 με 9 μέτρα ψηλότερη από σήμερα. Είμαστε περίπου στο 2100 ε, στις υποθέσεις μας και δεν ξέρουμε αν θα φτάσει η στάθμη της θάλασσας. 400 ppm διοξιδίου του άνθρακα είχαμε τότε και εάν δούμε τώρα τους παρόμοιους αριθμούς 405 διοξιδίου του άνθρακα, πέρσι τουλάχιστον, ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό συνέβαινε πριν από 3-5 εκατομμύρια χρόνια και η στάθμη της θάλασσας τότε ήταν πολύ ψηλότερη, 7 μέτρα τουλάχιστον ψηλότερη από τη σήμερα. Και για να έχετε και κάποιο σημείο αναφορά, η γη έχει πάγο μόνιμου πάγου στην Αντακτική και την Ακτική, που θα μπορούσε να αυξήσει κατά 7 μέτρα τη στάθμη τη θάλασσα παγκοσμίω, εάν έλειωναν. Ε, Βεβαίω, η Συμφωνία των Παρισίων δίνει ε, την αίσθηση ότι τα πράγματα είναι κατε... η ανάγκη είναι κατεπίγουσα να κάνουμε κάτι, αν θέλουμε να μείνουμε στον 1,5 βαθμό. Αλλά υπάρχει και αδράνεια στην κοινωνία. Υπάρχει παραλυσία στου πολιτικού και καμία δράση για την αλλαγή. Φαίνεται αυτό να είναι ένα κοινό σημείο μεταξύ πολλών διαφορετικών χωρών. Πρέπει να ε, βασιστούμε στα σφαιρικά μα συμπεράσματα από αυτή την έκθεση, ω προ το κατά πόσο είναι εφικτά κάποια πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι βάσει των νόμων τη χημία και τη φυσική είναι δυνατό να, παρα... να συγκρατήσουμε την υπερθέρμανση στον 1,5 βαθμό. Ναι, σε αυτό μπορούμε να βάλουμε τικ. Επίση έχουμε τα τεχνολογικά μέσα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μέτρα αναχέτησης και προσαρμογής και να γίνει ο κόσμος κάπως καλύτερος, ακόμη και αν είναι θερμότερος κατά 1,5 βαθμό. Ναι, είναι και αυτό εφικτό. Αν και πρέπει να γίνουν και άλλα τεχνολογικά βήματα. Ε, ανακατεύθυνση των ε, χρηματοοικονομικών ε, ροών συγκεκριμένα να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε τα ορυκτά καύσιμα, να τα επιδοτούμε. Αυτό είναι εφικτό. Ωστόσο, εκεί που υπάρχουν φραγμοί σήμερα είναι περισσότερο η χάραξη πολιτικής που δεν επιτρέπει να, μετα, να μεταλλαχθεί και να μετατραπεί η κοινωνία. Αυτό είναι το σημείο συμφόρησης όπου έχουμε κολλήσει και γι' αυτό τα πράγματα πάνε τόσο αργά και δεν μπορούμε να γίνουμε πιο φιλόδοξοι για να αναχαιτήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Πώς θα φτάσουμε λοιπόν τους στόχους μας. Για να περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη σε 1,5 βαθμό, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να μειωθούν γιατί για την ώρα αυξάνονται κιόλα, πρέπει να μειωθούν τα ερχόμενα 10 χρόνια. Μέχρι το 2030 πρέπει να μειωθούν κατά 45% σε σχέση μάλιστα με το 2010. 20% θα ήταν η μείωση για να περιοριστούμε στον 1,2 2 Για να, περιοριστούμε στον 1,5 βαθμό θα πρέπει να φτάσουν σχεδόν στο 0 εκπομπές διοξιδίου το 2050 σε σύγκριση με το 2075 ε, που θα ήταν το όριο για του 2 βαθμού. Θα πρέπει επίση να κοιτάξουμε και τι εκπομπέ που δεν είναι διοξιδίου του άνθρακα όπω το μεθάνιο από τη Γεωργία. Και αυτό θα είχε άμεσα ωφέλη για την ανθρωπότητα και τα ζωικά είδη. Να ολοκληρώσω με κάποια μηνύματα σε σημεία. Οι κλιματικέ αλλαγέ ήδη επηρεάζουν τι ζωέ των ανθρώπων, τα οικοσυστήματα και ε, την, ε, τη διαβίωση όλων ανά τον κόσμο. Εάν περιορίσουμε την υπερθέρμανση στον 1,5 βαθμό, θα έχουμε πετύχει κάτι το εφικτό, αλλά θα έπρεπε για να το πετύχουμε να δράσουμε αμέσω ε, με φιλοδοξία και για να κάνουμε αλλαγέ άνευ προηγουμένου σε όλη την κοινωνία. Υπάρχουν σαφή ωφέλη εάν διατηρήσουμε την υπερθέρμανση σε 1,5 βαθμό σε σύγκριση με του 2 ή περισσότερο, διότι κάθε μονάδα ή ε, κατοστιαία μονάδα ε, θερμοκρασία μετράει. Επίση, ο περιορισμό τη υπερθέρμανση 1,5 βαθμό πάει χέρι-χέρι με την επίτευξη και των υπόλοιπων στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μισό βαθμό λοιπόν μετράει. Κάθε παραπάνω βαθμό ζέστη μετράει. Κάθε χρονιά μετράει και κάθε επιλογή που κάνουμε μετράει. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much for your presentation, Professor. It uh, Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά για την παρουσίασή σας. Καλό τους συναδέρφους να πάρουν το λόγο για να ακούσουμε παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο catch the eye. Αν θέλετε το λόγο, παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σας. Ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Δείξατε στο τέλος της παρουσίασής σας σε ένα σκίτσο με τους πολιτικούς ε, που κρύβουν στην άμμο το κεφάλι τους. Παρακαλώ όμως εδώ να ε, ε, παρουσιάσετε περισσότερες αποχρώσεις. Ναι, εάν πάρουμε τον κύριο Τραμπ, ναι, αλλά είμαι πολύ περήφανος που πριν από κάποιους μήνες ο σύμβουλος του Προέδρου Ομπάμα είπε ότι χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχαμε συμφωνία για το κλίμα. Δεν είναι όλοι οι πολιτική από όλα τα μέρη του κόσμου ήδη. Σας παρακαλώ λοιπόν εδώ την επόμενη φορά στο θέμα αυτό να παρουσιάσετε περισσότερες αποχρώσεις. Επίσης, μια παρατήρηση σχετικά με τη δική σας τελευταία παρατήρηση. αυτή τη στιγμή με τον, ε, με τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο της Βραζιλίας που είναι ακόμη χειρότερος. Είναι δύσκολο να καταβάλουμε όλοι μαζί τις απαραίτητες προσπάθειες για να περιοριστούμε ε, σε αύξηση της θερμοκρασίας ε, στον 1,5 βαθμό. Όταν ε, συνάδελφοι ή κράτη-μέλη λένε ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε τίποτα αφού η Βραζιλία και οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν συμμετέχουν, παρόλα αυτά είναι απαραίτητο η Ευρώπη να καταβάλει προσπάθειες. Παρακαλώ να το σχολιάσετε αυτό. Να ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Χόισλινγκ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ναι, είναι ανησυχητικά τα στοιχεία. Και βλέπουμε την αποψήλωση των δασών στην Βραζιλία με την ευλογία του νέου Προέδρου. Είναι πολύ ανησυχητικό το ότι ακριβώς σε μια τόσο μεγάλη χώρα βλέπουμε να επιταχύνεται η καταστροφή των δασών. Η γεωργία λοιπόν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Αναφερθήκατε στα βιοκαύσιμα τα οποία αποτελούν τουλάχιστον ε, επίμαχο θέμα, διότι στην καλύτερη περίπτωση είναι ουδέτερα, στη χειρότερη περίπτωση είναι μάλλον επιβαρυντικός παράγοντας όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Με τεχνικά μέτρα φαίνεται να μην μπορούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις ε, και κάτι ακόμη μπορούμε με τις σωστές ε, γεωργικές μεθόδους ε, θα μπορέσουμε να μετριάσουμε την αλλαγή του κλίματος. Ε, όσον αφορά την παραγωγή κρέατος, ε, απαιτούνται πολλοί πόροι για την παραγωγή αυτή. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν και στον τομέα αυτόν. Και κάτι ακόμα το οποίο δεν αναφέρατε. Ως Ευρωπαίοι πολιτική πρέπει να κάνουμε πολλά, αλλά αν δούμε την ε, Γερμανία δεν πετυχαίνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Φέρουμε λοιπόν ευθύνη. Μπορεί πάντα να λέμε ότι υπάρχουν χειρότεροι από μας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φέρει τις ευθύνες της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκούτλαντ και κατόπιν θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για την ενδιαφέρουσα και σημαντική παρουσίασή σας και για την έκθεση που δημοσιεύτηκε τώρα το φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική έκθεση που είδαμε φέτος και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρη δεδομένη της διάσκεψης στο Κατοβίτσε. Λαμβάνουμε λοιπόν από εσά τις απαραίτητες πληροφορίες. Δύο παρατηρήσεις έχω δύο ενθαρρυντικά στοιχεία. Το ένα είναι η δική σας έκθεση και το άλλο θέμα είναι μια μαθήτρια στην Σουηδία που απήχε από το σχολείο της επί μήνες ε, λέγοντας στους ε, τοπικούς πολιτικούς ε, και σε άλλους πολιτικούς ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για το κλίμα. Το μήνυμά τη λοιπόν ήταν ότι έχουμε πια όλες τις πληροφορίες στη διάθεσή μα, τώρα πρέπει να δράσουμε. Και εσείς στην έκθεσή σα, μας λέτε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίσουμε, παρόλα αυτά θα θέσω κάποιε ερωτήσει. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεστε και δεν έχετε αναφέρει ακόμη, τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το, ο υπόλοιπος κόσμος όσον αφορά τα ποσοστά μείωση των εκπομπών, διότι το 2000, για το 2030 έχουμε τον στόχο μας του 40%. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι πρέπει να αυξήσουμε το στόχο αυτό στο 55%. Μήπως μπορείτε να το σχολιάσετε. Επίσης, έχω μια ερώτηση σχετικά με τα είδη ζώων που αναφέρατε και αναρωτιέμαι αν μπορείτε να μας πείτε τι ποσοστό ε, ζώων θα εξαφανιστούν εάν έχουμε αύξηση ε, της θερμοκρασίας κατά 1,5 και αύξηση θερμοκρασίας κατά 2% αντίστοιχα. Και τέλος, ε, μια ερώτηση σχετικά με τα δάση. Η χώρα μου, η Σουηδία, έχει πολλά δάση. Πώς πιστεύετε ότι μπορούν τα δάση να συνεισφέρουν και ως τόπος που δεσμεύει το διοξίδιο του άνθρακα, αλλά ε, και ως πρώτη ύλη. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> Thank you very much Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη εκ των προτέρων αν κάτι ξεχάσω. Πρώτα απ' όλα, για τους συναδέρφους από τη Γερμανία. Όχι, δεν θέλω να εκθέσω κανέναν μεμονωμένα εδώ σε αυτή την αίθουσα σε σχέση με την αδράνεια ή την άγνοια για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λαμβάνει υπόψη τα υψηλά επίπεδα φιλοδοξίας που χρειάζονται. Αλλά εμείς κάνουμε μία ανάλυση παγκοσμίω. Και όταν ε, ερχόμαστε να κάνουμε τέτοιες παρουσιάσεις, σας δίνουμε τη συνολική εικόνα. Είναι μια συνολική εικόνα, δεν πρόκειται μόνο για την Ευρώπη, οπότε Εννοείται ότι οι εξαιρούνται εξάλλου, όπως λέμε πάντα. Είναι σαφέ αυτό. Τώρα, για την βιοενέργεια. Και τι βιοενέργεια εννοούμε. Σίγουρα αυτή τη στιγμή εκμεταλλευόμαστε τον γεωργικό τομέα. Στη Βορεια Γερμανία από όπου έρχομαι εγώ το βλέπουμε πολύ εντατικά. Μάλιστα η κτηνοτροφία και η παραγωγή βιοαερίου είναι πράγματα που έχουμε πολύ εντατικά και τα επικρίνουμε. Στους υπολογισμούς αυτό που λαμβάνουμε υπόψη μας είναι τα δέντρα και τη χρήση της ξυλίας για την πρωτογενή ενέργεια και το διοξίδιο του άνθρακα το οποίο αποθηκεύεται τελικά είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε στην ε, προηγούμενη έκθεσή μας ως ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να μας επιτρέπει τον υπολογισμό των επιπτώσεων και το συναφές κόστος εξίας της ε, αλλαγής αυτής. Είναι καλό φυσικά να γίνεται μεγαλύτερη διαφοροποίηση, αλλά προς το παρόν αυτή είναι η εκτίμηση για την αφαίρεση του διοξιδίου του άνθρακα αμέσως, αφαιρώντας βέβαια την ενέργεια που περιλαμβάνεται στην γεωλογική αποθήκευση. Φυσικά και υπάρχουν ερωτήματα και φυσικά και υπάρχουν κίνδυνοι από την ίδια την αποθήκευση. Πρέπει να γίνει αποδεκτή αυτή η τεχνολογία και από το κοινό. Χρησιμοποιείται στην Νορβηγία η τεχνολογία αυτή, από όσο γνωρίζω, για το φυσικό αέριο που παίρνουμε από το διοξίδιο του άνθρακα. Η τεχνολογία αυτή υπάρχει και χρησιμοποιείται στη Βόρεια Θάλασσα. Που βέβαια είναι λιγότερο επικίνδυνο και για τον άνθρωπο αλλά σίγουρα υπάρχουν ερωτήματα και μια εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα είναι κάτι το οποίο ακόμα εξετάζουμε. Σα συμπέρασμα θα έλεγα αν μπορούμε να την αποφύγουμε, να την αποφύγουμε. Και έτσι έρχομαι στο δεύτερο σημείο σας που αναφερθήκατε στο οξύδιο του αζότου και στην παραγωγή κρέατος. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Και στην πρώτη έκθεση επίσης ε, συζητήσαμε για τους κλάδους αυτούς και τις συνέπειές τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Μεγάλη μείωση της κατανάλωσης του κρέατος αποτελεί ένα μέρος αλλαγής στην ανθρώπινη συμπεριφορά που είναι αναγκαίο. Δεν λέω ότι πρέπει να καταργηθεί πλήρω η κατανάλωση του κρέατος, αλλά σίγουρα να αποφύγουμε τη βιομηχανική παραγωγή κρέατος και την καθημερινή του κατανάλωση. Αν έχουμε 80-90% μείωση, αυτό θα βοηθούσε πολύ. Και οι μειώσεις αυτές, τα οξύδια του αζότου, που συνδέονται με την κτηνοτροφία ακριβώς, είναι επίσης κάτι σημαντικό γιατί όσο περισσότερο μειώνουμε το διοξίδιο του άνθρακα, τόσο περισσότερο θα επηρεάζουν τα οξύδια αυτά τη διαμόρφωση του κλίματος στο μέλλον. Άρα είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Γιατί είναι επίσης αέρια του θερμοκηπίου, δεν είναι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτή, οι λοιπόν εξετάζονται και για να έρθω τώρα στην ερώτηση της Σουηδέζας, απάντησα κάπως στην ερώτησή σας για τα δάση και τη χρήση τους. Η ανάκαμψη των δασών θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα σε συνδυασμό με τον περιορισμό των εκπομπών για να εποφεληθούμε περισσότερο από τη διατήρηση της βιοπικιλότητας, τρόφιμα για όλους, διατήρηση των οικοσυστημάτων και έχοντας στη διάθεσή μας αρκετές περιοχές όπου να προστατεύεται η βιοπικιλότητα. Όλα αυτά είναι και ωφέλη για το κλίμα, οπότε τι να κάνουμε. Αυτό το οποίο χρειάζεται, και εγώ δεν είμαι πολιτικός, έτσι, αλλά μελετώντας το έργο των ε, πολιτικών έχω καταλήξει σε αυτό, ότι οι πολιτικοί θα έπρεπε να συμφωνήσουν μεταξύ τους για μεγάλες κλίμακας αλλαγές που να καλύπτουν μεγάλες επικράτειες, όχι μόνο να κρυβίνουν εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά να μειωθεί και η τιμή των προϊόντων τα οποία παράγονται με βιώσιμο τρόπο, τα βιολογικά προϊόντα ας πούμε να είναι προσιτά για όλους. Και ό,τι προέρχεται από τη βιομηχανική γεωργία και εκτινοτροφία να κρυβίνει για να υπολογιστεί στην παραγωγή αυτή και το κόστος της καταστροφής στο περιβάλλον. Η διεθνής αυτή συνεργασία όμως που απαιτείται, και έτσι έρχομαι σε ερώτημα του πρώτου ομιλητή, διεθνή συνεργασία είναι προϋπόθεση και αυτό είναι ένα στοιχείο αδράνειας των πολιτικών που ανέφερα. Τώρα για τους ε, στόχους για το κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1,5-45% μείωση σε σχέση με το 2010. Όμως για όλους εμάς το σημείο αναφοράς είναι το 1990. Αν πάρουμε λοιπόν την αξία για το 1990 για την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε μείωση κατά 15% σε σχέση με το 2010. <laughs> Και για να πετύχουμε την μείωση κατά μέσο όρο που χρειάζεται, χρειάζεται περισσότερο. Αυτό μου σημαίνει ότι όλοι πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κάνουν το ίδιο. Όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε διεθνές επίπεδο οι ε, αναπτυσσόμενες χώρες έχουν διεκδικήσει ε, περισσότερο τη χρήση στερεών καυσίμων από ότι ο δυτικός κόσμος, ε, Τουρκία, στην Αφρική χώρες θέλουν την ε, βιομηχανία. Όμως, όσο λιγότερα κάνουν αυτές οι χώρες, τόσο περισσότερο πρέπει να κάνουν οι βιομηχανοποιημένες οι χώρες για να πετύχουν το στόχο μας. Έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας για τη θνησιμότητα. Δεν μπορώ να σας δώσω τα νούμερα όσον αφορά τον κίνδυνο θανάτου ε, για τα ζώα. Αυτό όμως που γνωρίζουμε από την επιστήμη είναι ότι όλες αυτές οι αρχές σχετικά με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας που ισχύουν για τον άνθρωπο ισχύουν και για όλα τα θηλαστικά. Βέβαια κάποια αντέχουν περισσότερο, κάποια κάπως λιγότερο. Πάντως υπάρχουν επιστημονικές εκθέσεις για ε, την άνοδο της θερμοκρασίας και την παραγωγικότητα στα ζώα και πως αυτή επηρεάζει την ε, παραγωγικότητά τους. Και άρα, αν δεν υπάρχει μάλιστα και αρκετό νερό, καταλαβαίνετε ότι σαφώς και θα υπάρξει αύξηση στην θνησιμότητα ε, των ε, κοπαδιών. Το ίδιο ισχύει για μας. Δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι θα χάνουν τη ζωή τους ε, περισσότεροι από ό,τι σήμερα, αν δεν περιορίσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας. Ήδη από το 2003 το ξέρουμε. Εκεί υπήρξε στην Ευρώπη κύμα καύσωνα και το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει προσαρμογή σε τέτοια φαινόμενα. και πάντα οι πιο ευάλωτοι, οι πιο φτωχοί, αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά στις ε, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εκτίθενται περισσότερο και αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο βέβαια. Σε κάποια σημεία του πλανήτη δεν θα μπορούν πλέον να κατοικήσουν άνθρωποι ακριβώ ακριβώς αυτής της κλιματικής αλλαγής. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Άλλε ερωτήσει τώρα. Κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Πραγματικά ήταν ε, πολύ κατατοπιστική αυτή η πληροφόρηση και η διαφοροποίηση που κάνατε μεταξύ του 1,5 βαθμού και των 2. Το πακέτο ενέργεια και κλίμα που ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο για την Ενεργειακή Ένωση με τους στόχους που θέσαμε 32% ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως το 2030, 32,5% αποδοτικότητα και 40% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου είναι ένα πρώτο βήμα. Εδώ θελήσαμε να καταρτήσουμε μια μακρόπνοη στρατηγική. Την Τετάρτη ο Επιτροπός μας θα παρουσιάσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική ο οποίος έχει ε, θέσει στόχο τον 1,5 βαθμό. Έχουμε πει όμω μηδενική εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα έω το 2050 και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εσεί πώ το βλέπετε, πώ βλέπετε ότι μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Διότι οι μηδενικέ εκπομπέ μέχρι το 2050 είναι εφικτό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια μετατόπιση τη χρήση τη ενέργεια ω το 2040. Και επίση η στρατηγική μα για το μεθάνιο ήταν αρκετά δυναμική και είναι σαφές ότι σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα το μεθάνιο συμβάλλει περισσότερο στην ε, αύξηση του, της ποσότητας των αερίων του θερμοκηπίου. Ήθελα λοιπόν αυτό να το δούμε προσεκτικά. Σήμερα στην Μοντ, τι διαβάζω, οι γαλλικές τράπεζες χρηματοδοτούν το πετρέλαιο και τον άνθρακα με μεγάλα ποσά. Οι γαλλικές τράπεζες ε, ε, αφιέρωσαν 71% των χρηματοδοτήσεων τους στα ορυκτά καύσιμα. Δεν θα ήταν λίγο ενδιαφέρον να κοιτάξουμε τι κάνουν και οι τράπεζε, διότι αν οι τράπεζε χρηματοδοτούν την καλλιέργεια τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, θέλουμε ο κόσμο να ε, πάρει μέρο σε όλη αυτή την προσπάθεια και μετά βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Ε, ο κόσμο αρνείται τι αλλαγέ, βλέπετε τι έγινε με τον ντίζελ και τα αυτοκίνητα και λέει τι κάνουν οι κυβερνήσει, τι κάνουν οι τράπεζε και δεν θέλουμε να πληρώνουμε φόρου. Ε, αυτό συμβαίνει στο τέλο. Πρέπει να πληροφορούμε του πολίτε, αλλά θα πρέπει και η πολιτική να είναι υποδειγματική. Ε, πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, διότι σε αυτό το πλανητικό χωριό πρέπει να έχουμε μια συμπεριφορά υποδειγματική όλοι. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Χερμπράντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ καθηγητά που ήρθατε εδώ για να παρουσιάσετε τα πορίσματά σας και τις σκέψεις σας. Είναι πολύ θετικό που είχατε τόσο να μας πείτε. Το μήνυμά σας φαίνεται κάπως απεσιόδοξο, ε, λίγο ζωφερό, αλλά και υπάρχει μια ελπίδα, μια χτίδα φωτός. Δηλαδή ότι μπορεί κάτι να γίνει αν μείνουμε στον 1,5 βαθμό και δεν φτάσουμε στους 2. Αλλά υπό την θα πραγματοποιηθεί αυτό. Το είδα στις διαφάνειές σας ε, πραγματικά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η κοινωνία δεν είναι ακόμα έτοιμη για τις ριζοσπαστικές αλλαγές που χρειάζονται για να μείνουμε κάτω από τον 1,5 βαθμό. Αν και είναι απαραίτητο αν ακούσει κανείς την παρουσίασή σας. Νομίζω το γαλλικό παράδειγμα ε, αναδεικνύει ανά, ε, ανάγλυφα αυτό που λέτε. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης λόγω των κλιματικών αλλαγών είναι ήδη Κάτι που πυροδοτεί διαμαρτυρίες σε επίπεδο κοινωνίας. Έχω τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η μία είναι η δήλωσή σας ότι από τεχνολογικής σκοπιάς είναι εφικτό να μείνουμε μέσα στα όρια του 1,5 βαθμού ή κάτω είχα την αίσθηση ότι δεν αναφερέωσαστε μόνο σε μελλοντικέ ε, τεχνολογικές φοβερές ριζοσπαστικές λύσεις, αλλά αναφέρατε και πολλές τεχνολογικές λύσεις που ήδη είναι διαθέσιμες. Μπορείτε να το αναλύσετε. Χρειαζόμαστε εφευρέσεις, καινούριε. Πόσες. Και η άλλη μου ερώτηση αφορά τη βιοπικιλότητα. Το, καν... το καταστήσατε σαφές με του κορυκλογενείς υφάλους και την ε, βιολογική ενέργεια και την ε, αποθήκευση και κράτηση του άνθρακα. Κάνουμε τα οικοσυστήματα ιδιαίτερα ευάλωτα. Αλλά μπορείτε να μας πείτε περισσότερα στοιχεία, αν κινηθούμε προς τον 1,5 βαθμό, τι προσδοκίες υπάρχουν ως προς την βιοποικιλότητα και την απώλεια ζωικών ειδών. Και η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με αυτό το λίγο σκοτεινό που αναφέρεται, την κρίζα ζώνη, το σημείο που υπάρχει η αλλαγή, ε, το κρίσιμο σημείο. Σίγουρα εκεί, εάν περάσουμε το κρίσιμο σημείο, δεν θα μπορούμε καθόλου να ελέγξουμε το κλίμα. Θα έχει ξεφύγει από τον ελεγχό μα η όλη κατάσταση. Αλλά με ανησύχησε πολύ αυτό που αναφέρεται με τι τρελέ θερμοκρασίε ε, για το καλοκαίρι που πέρασε. Και πριν από λίγε εβδομάδε στην Αρκτική κιόλα. Έχετε την εντύπωση ότι ήδη μάλλον στην Αρκτική είμαστε σε αυτό το κρίσιμο σημείο ή δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από τα μοντέλα που έχετε χρησιμοποιήσει στην έρευνά σας. Ευχαριστούμε κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ καθηγητά. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση και μια ερώτηση και σε σχέση με την ανακοίνωση για την ε, ε, υπερθέρμανση του πλανήτη και τις κλιματικές αλλαγές. Εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθειά σα να αντιστρέψετε το μήνυμα μιλώντα για τα ωφέλη του να παραμένουμε στον 1,5 βαθμό και να αντί να επιμείνετε στα μειονεκτήματα των προβλέψεων των 2 βαθμών. Όμω, εάν συγκρίνουμε τα σενάρια του 1,5 βαθμού με του 2, φαίνεται ότι απέχουμε από την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτε. Ήδη με τον 1 βαθμό πάνω από το όριο, το σημείο αναφορά δηλαδή, της βιομηχανικής εποχής έχουμε θανάτους, καταστροφές και τεράστιες οικονομικές ζημιές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν χειροπιαστοί απτοί λόγοι. Το βιώνουν ήδη οι πολίτες στη ζωή τους. Δεν συμμερίζομαι την επικοινωνιακή σας απόπειρα που μας πάει στην προϊστορία. Το 2100 θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος που ήδη ελπίζει στις μολυπτικέ γενέ και θέλουμε να τους εξασφαλίσουμε ένα καλό μέλλον. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Τώρα άλλο είναι να μιλάμε για μακρινές εποχές. Πρέπει να σκεφτούμε τι συμβαίνει ήδη στην Αρκτική, στους οι υφάλους, αλλά όχι μόνο στις μακρινές περιοχές. Δίπλα μας, πλημμύρες, ε, ε οι κατολιστήσεις, οι καταιγίδε ξαφνικές. Αυτό είναι που πρέπει να μα απασχολήσει και για την τεχνολογία. Ε, μην επιμένουμε μόνο στι τεχνολογικέ λύσει. Δεν θα είναι υπεύθυνοι τη τεχνολογία που θα φέρουν την ε, θεραπεία στο πρόβλημα, διότι αυτοί κοιτάνε μόνο το οικονομικό κέρδο. Οπότε, ήθελα να μου πείτε, το πρόβλημα είναι η επιστημονική μονανάλυση των συνεπειών τη υπερθέρμανση του πλανήτη, μήπω πρέπει να ασχοληθούμε με το γεγονό ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμο, οι πολίτε, οι λαοί, ότι υπάρχουν χειροπιαστέ συνέπειε από τις κλιματικές αλλαγές. Ο κόσμος πληρώνει τις συνέπειε τώρα, όχι αυτοί που θα ζουν το 2100. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Θέλει άλλο κάνει το λόγο. Εάν όχι, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια σειρά πολύ καλών ερωτήσεων. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την ερώτηση για τη μείωση των εκπομπών. Εάν πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει ουδέτερη ως προς τις εκπομπές μέχρι το 2040, αυτό θα ήταν πολύ ενθαρρυντικό, αλλά δεν μπορώ να σας πω εγώ σε τι βαθμό αυτό είναι ρεαλιστικό στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, διότι δεν έχω αρκετές πληροφορίες στα χέρια μου αναφερθήκατε σε ένα από τα βασικά εμπόδια που είναι η χρηματοδότηση, η επιδότηση των ε, ορυκτών καυσίμων, κάτι που βλέπουμε ακόμη, ιδιαίτερα όσον αφορά τον άνθρακα και τα θερμοελεκτρικά εργοστάσια. Αυτό λοιπόν είναι καταστροφικό για το κλίμα. Διαιωνίζεται έτσι μια τεχνολογία που θα μας δυσκολέψει πολύ ε, στην ε, αναχέτηση της αλλαγής του κλίματος, ε, διότι μέχρι το 2050 και σύμφωνα με το στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, Ε, κάθε εκπομπή που πραγματοποιείται σε ένα μέρος ε, θα πρέπει να αντισταθμιστεί σε άλλον τομέα. Και οι αερομεταφορές και η ναυτιλία είναι σημαντική προβληματική τομής όπου απαιτούνται Βελτιώσει στην τεχνολογία και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιες βασικές αρχές ε, για να ε, βρούμε υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το εξής ε, και στη Γερμανία τα ίδια ισχυρίστηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Η αύξηση των των τελών ε, στο ντίζελ και τη βενζίνη είναι ένα πρώτο μέτρο το οποίο όμως ε, κάνει τους ανθρώπους ε, να δυσανασχετούν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε το κόστος και ιδιαίτερα όχι στους στοχούς και στις ευάλωτες ομάδες των πολιτών μας. Αυτό λοιπόν είναι πολιτικό καθήκον, ε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να επιληθεί για να αποφύγουμε τη δυσαρέσκεια των ανθρώπων. Όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνολογιών, νομίζω ότι το βασικό θέμα είναι ότι για κάποιες από τις τεχνολογίες ε, πρέπει να πετύχουμε τον στόχο όσον αφορά τη διάδοση της χρήσης τους. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, τα συνθετικά καύσιμα, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην αυτιλία και στις αερομεταφορές. Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει πολύ περισσότερες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ε, ηλιακή και αιωλική, καθώς ε, και η τεχνολογία του υδρογόνου. διότι ακόμη βλέπουμε χρήση μεθανίου κυροζίνης στην αυτιλία. Υπάρχουν ε, λοιπόν δυνατότητες. Βλέπουμε να χρησιμοποιούνται σε περιορισμένο βαθμό κάποιες τεχνολογίες. Εγώ οδηγώ με χρήση φυσικού αερίου και μάλιστα με ανακύκλωση των ε, αερίων. Χρειάζεται λοιπόν επένδυση στα διζελοκίνητα οχήματα. Και χρειάζεται αντικατάσταση της τεχνολογίας όταν ε, οι πολίτες αντικαθιστούν ούτως ή άλλως τα παλιά τους ε, οχήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια όθηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κάτι τέτοιο σίγουρα θα ήταν πολύ καλό. Χρειαζόμαστε λοιπόν εναλλακτικέ πηγές ενέργειας. Πρέπει να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση. Και έτσι θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε εναλλακτικέ ε, μορφές ενέργειας στις μεταφορές. Και ίσως θα έπρεπε να έχουμε μια μεταβατική περίοδο, αντί απλά να αυξάνουμε τη φορολογία στο ντίζελ και τα άλλα καύσιμα. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να έχουμε δωρεάν δημόσιες μεταφορές και να έχουμε σημαντικές ε, επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Ο στόχος του 1,5 βαθμού αναφέρεται στις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για να πετύχουμε μια τέτοια τεχνολογική μετάβαση. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ θα χρειαστούν για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Για να πετύχουμε τον απαραίτητο μετασχηματισμό. Κάποιοι μάλιστα έχουν συγκρίνει αυτόν τον μετασχηματισμό με τον μεταπολεμικό μετασχηματισμό. Είναι λοιπόν, νομίζω, σημαντική προϋπόθεση το να εγκαταλείψουμε τις παλιές τεχνολογίες. Όσον αφορά το θέμα της βιοπικιλότητας, στην τελευταία έκθεση αξιολόγησης δεν καταφέραμε να ε, εντοπίσουμε κάποιο είδος που να έχει εξαφανιστεί λόγω της αλλαγής του κλίματος. Τώρα νομίζω ότι αναφέρεται ένα είδος που είχε εξαφανιστεί, αλλά συνδυασμός παραγόντων οδηγεί σε μείωση της βιοπικιλότητας. Και βλέπουμε βιο και βλέπουμε απώλεια της βιοπικιλότητας σε κάποιες περιοχές, ε, στις ε, τροπικές ζώνες. Ε, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται τα ίδια αυτά, σημαίνει ότι χάνουν τους φυσικούς οικότοπούς τους. Θα συμφωνούσα με τον με τον όρο μαζική εξαφάνιση, η απώλεια τροπικών ειδών έχει διαπιστωθεί και η παρούσα εξαφάνιση είναι η μεγαλύτερη που είδαμε τα τελευταία 50 εάν όχι 300 εκατομμύρια χρόνια. Η αλλαγή του κλίματος, λοιπόν, έχει καταστροφικές συνέπειες. Και είναι επίγον να μετριάσουμε την αλλαγή του κλίματος. Υπάρχει και το θέμα της επικοινωνίας, της ενημέρωσης. Σίγουρα Βλέπουμε αντίκτυπο στην Ευρώπη, βλέπουμε ακραία φαινόμενα και στην IPCC. Μιλάμε για αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης ακραίων φαινομένων. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο στατιστικά και μεθοδολογικά να αποδώσουμε ένα συγκεκριμένο φαινόμενο στην αλλαγή του κλίματος. Είδαμε τις πλημμύρες στην Ιταλία, είδαμε την ξηρασία του περασμένου καλοκαιριού και σίγουρα κρούν τον κόδωνα για όποιον ενδιαφέρεται για τον τομέα αυτό, αλλά το να πούμε ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο στο συγκεκριμένο μέρος ε, οφείλεται στην αλλαγή του κλίματος είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ισχυριστούμε. Αυτό όμως που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτά που παρατηρούμε ευθυγραμμίζονται με τις προβλέψεις της IPCC τα τελευταία 30 χρόνια. Ευθυγραμμίζονται λοιπόν με τις προβλέψεις αυτές και μπορεί αυτή τη στιγμή να τα θεωρούμε ακραία φαινόμενα, αλλά σε 30-40 χρόνια θα είναι πια ο κανόνας. Αυτό λοιπόν είναι μια πτυχή που πρέπει να τονίσουμε. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ε, η αλλαγή του κλίματος κατά 1,5, η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό Κελσίου σίγουρα είναι καλύτερο από αύξηση κατά 2 βαθμούς Κελσίου, διότι η αύξηση κατά 2 βαθμούς Κελσίου θα σημαίνει ότι θα ζούμε σαν έναν τελείως διαφορετικό κόσμο και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη στο πλαίσιο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, κύριε Πόρτνερ. Πολύ μας βοήθησε και ιδίως σε σχέση με την διάσκεψη του Κατσοβίτσεκ. Ευχαριστούμε πολύ. Uh, Ωραία, λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε, περνάμε σε ένα ψήφισμα που έχουμε για τα νότατα επίπεδα διαφόρων ε, ουσιών σε διάφορα προϊόντα αμυντοσουλφουρίν, μπιφενόξο, κλωριπυρός, κλωριπυρός κτλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι συνεισηγήτρια, οπότε πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τους συναδέρφους που βοήθησαν στην εκπόνηση του ψηφίσματος αυτού, λέει η κυρία Κοντίν. Πρόκειται για την αναθεώρηση προς τα πάνω ανώτατων ορίων υπολείπων από το σημαντικό στα... στις ελιές, τις επιτραπέζιες ελιές και στην παραγωγή του λαδιού. Προτείνει το LMR για την ελιά να τριπλησιαστεί και από 0,9 μιλιγκράμμα ανά κιλό να πάει σε 3 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Ε, πραγματικά πρόκειται για ε, μια μεταχείριση επί 4 σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν βασίζεται σε μελέτη της ΕΦΣΑ που λέει να μειωθούν οι τιμές για όλα τα αγροτικά προϊόντα, συγχρόνως όμως να αυξηθούν για την ε, ελιά. και και καλή. Οι συστάσεις αυτές έρχονται μετά από την ε, σημαντική κρίση που έχουμε στην Νότια Ευρώπη από το 2013 που έχει να κάνει με το φαστιζιόζα που είναι βακτηρίδιο το οποίο πλήττει την περιοχή εδώ και καιρό. Και αυτό επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι μέσα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, γιατί τα διάφορα πρωτόκολλα για τη μη διάδοση της ε, αρρώστιας επέτρεψαν το ασημιπρίτ, που είναι ένα κοτινοειδές, να χρησιμοποιηθεί ευρέως, ενώ στη Γαλλία απαγορεύεται. Και τρίτον, επειδή η πρώτη αύξηση των ανώτατων επιπέδων υπολείπου το 2016, ε, που έγινε το 2016, τώρα η Επιτροπή θέλει να πολλαπλασιάσουμε επί τρία τα επιτρεπόμενα επίπεδα. Δεν πρέπει όμως να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η πραγματικότητα είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλος όγκος προϊόντων τέτοιων και πρέπει να διατεθούν. Όμως υπάρχει μελέτη αντικτύπου και το σιταμιπρίτ είναι ένα προϊόν το οποίο σκοτώνει της ε, μέλισσας και από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο χρησιμοποιείται όταν ακριβώς ε, οι μέλισσες δραστηριοποιούνται πολύ. Πρόκειται έτσι καλλιώς για εντατικοποίηση, οπότε οι επιπτώσεις στο θάνατο τους επικονιαστές είναι πολύ επικίνδυνο για τους επικονιαστές λοιπόν, γιατί κινδυνεύουν με θάνατο. Υπάρχουν εναλλακτικέ στο Snapdragon όμως που θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε έτσι καλύτερα τις ελιές, αλλά υπάρχουν και άλλες θεραπείες. Υπάρχουν τα αποτελέσματα του Πανεπιστήμιου του Σαλάντο στην Ιταλία με πολύ καλά αποτελέσματα Και από την άλλη, προκειμένου να πετύχουμε τους κατά προτεραιότητα στόχους μας, δηλαδή την προστασία της υγείας, μια στιγμή γιατί χάθηκα λίγο, λέει ο Μιλήτρια. Είναι δυνατόν, χάρη στην καινοτομία, χάρη στην ανάληψη ευθύνης, και δεδομένου ότι έχουμε διάφορες αντιφατικές ε, απόψεις, στο δεύτερο παράρτημα έχουμε προσθέσει μια πιο συνεπή πρόταση για την ελιά. Η Επιτροπή στις διάφορες ε, μελέτης της ε, διαμαρτύρεται για τη μείωση των επικοινωνιαστών. Ναι, αλλά τότε οι προτάσεις της θα πρέπει να είναι συνεπείς με την ανησυχία αυτή και άρα να χρησιμοποιούνται παρασιτοκτόνα που να είναι πιο βιώσιμα και που να μην καταστρέφουν. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς βάζουμε προτεραιότητα την προστασία της υγείας και της βιοπικιλότητας. Γι' αυτό σας παρακαλώ να υποστηρίξετε την αντίρρηση αυτή, την ένστασή μας αυτή. Ευχαριστούμε εκ μέρους του κύριου Πάλλας, η κυρία Κάντενμπαχ. ein herzliches Dankeschön. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του συναδέλφου Πάλλας. Όσον αφορά λοιπόν ε, την ε, τα στις ελιές πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρόκειται για νεονικοτινοειδές ε, το οποίο χρησιμοποιείται ως εντομοκτόνο. Όπως και οι άλλες ουσίες που απαγόρευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχές του έτους η ακεταμιπρίδη ε, θέτει σε κίνδυνο τους ε, επικονιαστές ε, και δημιουργεί και άλλου κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν πρότεινε συνέχιση της απαγόρευση. Αντιθέτω, επιτρέπει τριπλάσια κατάλοιπα στο ελαιόλαδο, ενώ αρχικά είχαμε 0,09 μιλιγκράμμ ανά κιλό, τώρα έχουμε 3 γραμμάρια ανά κιλό. Το 2016 επιτρεπόταν 0,1 ε, μιλιγκράμμ, το οποίο αυξήθηκε τότε στα 0,9 και Αυτό δείχνει ε, την ε, αύξηση της χρήσης της σε κάτι που οδηγεί σε επιπτώσεις και για τους ανθρώπους και για τα ε, έντομα. Το 80% ε, των εντόμων στην Ευρώπη έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια και απειλούνται από μαζική εξαφάνιση. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τον τρόπο ε, που, καλλιέργειας και να απαγορεύσουμε τις ουσίες αυτές υπάρχουν και κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Στην ε, γνωμοδότηση η ΕΦΣΑ δεν λαμβάνει υπόψη της αυτό το ε, cocktail effect, ε, της επιπτώσεις από την συνδυασμένη χρήση διαφόρων ουσιών Ε, πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας για να καταλάβουμε τι συνέπειες έχουν οι ουσίες αυτές στην ανθρώπινη υγεία και έτσι πρέπει να εξετάσουμε το θέμα γενικότερα και όχι μόνο να εξετάσουμε το επίπεδο καταλήπων στις ελιές. Θα πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τους πολίτες μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν βιώσιμη και ολοκληρωμένη προσέγγιση και υπάρχουν ήδη εναλλακτικέ τεχνικές για να προλάβουμε τη ζημιά στις καλλιέργειες και να προστατεύσουμε τα φυτά. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να προσφέρουμε ε, βιώσιμες λύσεις στους γεωργούς. Η χρήση της ακεταμιβρίδης ε, ε, δεν συνάδει με, την, με τους στόχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προστατεύσει το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξανασκεφτεί τη θέση της και να μειώσει τα όρια για την ακεταμιπρίδη στα 0,5 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε η κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ τα ίδια επιχειρήματα έχω όπως και οι συνάδελφοι. Ίσως θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε ότι είναι η μόνιμη επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανατίθενται τα θέματα των φυτών, η Σκοπάφη, η οποία ενέκρινε ε, ένα ανώτατο επίπεδο και εξού και ένστασή μας γιατί δεν είναι δυνατόν. Απ' τη μια πρόκειται για το νοικοτοειδή και ξέρετε ότι τα απαγορεύουν χώρες όπως η Γαλλία και έτσι κι γενικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα μειώνουμε όσο μπορούμε σε όλα τα απορροκυπευτικά. Η πρόταση όμως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα αυξάνει. Μάλλον τα μειώνει παντού εκτός από το λάδι, το ελαιόλαδο και την ελιά. Και τι σημαίνει αυτό, ότι θα σκοτώσουμε τις μέλισσες, τους επικονιαστές, θα σκοτώσουμε τέντονα, γιατί τα νεονικοτοειδή δεν ξεχωρίζει οι μέλισσες και τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα είναι η ξύλα της που είναι ένα βακτηρίδιο, στη Νότια Ιταλία. Να, μα Ιταλή. Και στην Κορσική βέβαια και στη Νότια Γαλλία το έχουμε. Και τι λένε, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το παρασιτοκτόνο, το οποίο όμως θα έχει επιπτώσεις και στην υγεία και στη βιοποικιλότητα, αλλά και την υγεία. Γιατί όσο περισσότερο θα επεκταθεί το προϊόν αυτό, τόσο περισσότερο θα επικεντρώνεται στο λάδι. Και όταν κοιτάζω τα νούμερα, τι βλέπω ότι ήδη το 2016, και το είπε και συνάδελφος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη αυξήσει επί 3, ήταν 0,01 και πήγε στο 0,09 και τώρα θέλουμε να πάει σε 3 μιλιγκράμμ ανά αυτό σημαίνει ότι επί 10 και επί 20 θα ψεκάζουμε. Υπάρχει Επιτροπή για τα Παρασιτοκτόνα και βλέπουμε και την κινητοποίηση των πολιτών που δεν θέλουν πια τοξικά παρασιτοκτόνα που έχουν ευαισθητοποιηθεί με την απώλεια της βιοπικιλότητας. Οπότε δεν βλέπω, αφού υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις, γιατί να αυξήσουμε το LMR. Στέλνω μήνυμα λοιπόν προς όλους τους συναδέρφους. Αύριο θα ψηφίσουμε και πρέπει να ψηφίσουμε αυτή την ένσταση. Κάναμε μια πρόταση, υπάρχει ο κατάλογος, ε, θέλουμε 0,5 και δεν θέλουμε ελιές που να παράγονται με αυτό το παρασιτοκτόνο. Για τελειώς όλοι θα ψωνίζουμε βιολογικά προϊόντα. Όταν βλέπετε από την Ιταλία λάδι, πάντα θα σκέφτεστε ότι αφού αυξήσαμε το ελεμέρ, προφανώς θα υπάρχει μέσα σε αυτό το λάδι. Οπότε καλύτερα να μην παίρνω αυτό το λάδι, να παίρνω κάτι άλλο είτε με λιγότερη συγκέντρωση ιδεολογικό. Εξού και πρέπει να έρθετε να ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Θα δούμε τι θα γίνει με τις ηλιές. Η Σκιώδης τώρα. Ο κύριος Τουρκάνο ήταν, αλλά τον αντικαθιστά εδώ ο συνάδελφος. Παρακαλώ, κύριε Χάντσα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, ζητώ συγγνώμη που δεν εδώ ο συνάδελφος μου ζήτησε να διαβάσω αυτά που θα έλεγε. Στόχος του σχεδίου ρύθμισης της Επιτροπής ε, ζητάει να μειώσουν τα ανώτατα επίπεδα για διάφορα ε, και την ακετοκομπρίνη και τα λοιπά και προτείνει αύξηση ...τον τιμών στις επιτραπέζιες ελιές και το λάδι. Ε, βρώμη και λοιπά για προϊόντα που περιλαμβάνουν ακέτομη πυρίδι. Στην αξιολόγηση κινδύνου με χώρες όπως η Πολωνία και η Ιταλία η ΕΦΣΑ είπε ότι είναι ασφαλή τα όρια αυτά για τους καταναλωτές. Εμείς γνωρίζουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει η προστασία των πολιτών, αλλά πρέπει να αναφέρουμε ότι η ρύθμιση θέλει να καλύψει διάφορα προϊόντα. Δεν έχουν εντοπιστεί από την ΕΦΣΑ ε, κίνδυνοι στις ε, δοκιμές που έγιναν όσον αφορά την ακετά μυπρίδη. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία. Και μάλιστα με τις τρέχουσες τιμές 0,9 μιλιγκράμμα ανά κιλό θεωρείται μια καλή πρακτική. Είναι τιμές που εγκρίθηκαν το 2016. Συνεπώς και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ε, τις ασθένειες οι οποίες έχουν προκύψει στην Νότια Ευρώπη χρειάζεται το χρέστη ουσία αυτή. Με 0,5 δεν μπορούμε να έχουμε ουσία με τέτοια περιεκτικότητα που να μπορεί να καταπολεμήσει την ασθένεια. Η πρόταση επιτροπής ευθυγραμμίζεται πλήρως και με τον κανονισμό 396 του 2005, σημείο 14.1, λαμβάνει υπόψη της όλες τις ισχύουσες μέχρι τώρα ρυθμίσεις για τα παριστοκτόνα. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Hansen. Now, Mr. Pedicini. Ευχαριστούμε, κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα. Θέλω να πω Θέλω να καθησυχάσω αυτούς που συνυπογράφουν αυτή την πρόταση, την ένσταση. Τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια τη ουσία αυτή. Διότι το γεγονό ότι χρησιμοποιείται μαζικό στην Ιταλία για την καταπολέμηση τη ξυλέλα φαστιντιόζα δεν σημαίνει ότι εμεί θέλουμε να χρησιμοποιείται. Την απόφαση αυτή δεν πήρε ο Πρωθυπουργό. Είμαστε αντίθετοι στην ε, συστηματική χρήση αυτών των ε, φυτοκτόνων, των ζυζανιοκτόνων μάλλον. Θα έπρεπε να υπάρχει επιλεκτική εκρίζωση. Φυτογενομικά βιώσιμα μέτρα όπως ε, η αγωγή για τα φυτά. Όμως την Ιταλική κυβέρνηση τώρα κυβερνούν ε, επικίνδυνοι λαϊκιστές, ε, λένε. Και τώρα βλέπετε πως αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Εγώ λοιπόν στηρίζω την ένσταση. Η κυρία Γκαρντίνη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς ως Ιταλία και ως Ιταλική πραγματικότητα και σύστημα και Ιταλική αντιπροσωπεία κιόλα. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ε, ε, υπερψηφίσουμε αυτή την ένσταση, διότι θα ψηφιζόταν εάν υπήρχε η απόρριψη αυτή τη αύξηση των μεγίστων επιτρεπωμένων ορίων. Ακόμη και αν η Επιτροπή αποδεχόταν την ε, γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ που κατέληξε ότι δεν υπήρχαν ε, κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, τους καταναλωτές, και επειδή πρόκειται για ένα νεονικοτινοειδές, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία των μελισσών, Θεωρούμε ότι μπορούμε να δεχτούμε μια ε, θέση που βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης, της πρόληψης. Η ένσταση θέλει να μειώσει τα επιτρεπόμενα όρια του ζυζανιοκτώνου. 0,5 μιλιγκράμμ ανά κιλό αντί 0,9 που ισχύει τώρα. Πραγματικά ε, εκπλήσωμαι όταν ακούω τέτοιες επιθέσεις προς έναν οργανισμό, ευρωπαϊκό κιόλας οργανισμό, ευρωπαϊκή αρχή, όπως η ΕΦΣΑ, με λόγια που βρίσκω αρκετά ανησυχητικά κιόλας. Ε. Δηλαδή θα μπορούσε κανείς, κατά την άποψή μου, ε, τελείως θεμητό είναι, να μην συμφωνεί με την άποψη κάποιου, αλλά μπορεί να προβάλλει αντεπιχειρήματα Τώρα να πηγαίνει να αμφισβητεί το κύρος ε, της ΕΦΣΑ, ναι. της αρχής αυτής, ε, λίγο ξεπερνάει τα όρια. Ξεπερνάει την ε, θεσμική κοσμιότητα, για να το πω έτσι. Ο καθένας βέβαια είναι υπεύθυνο για τα δικά του τα λόγια, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να σημειώνονται και να τα παίρνουμε σοβαρά υπόψη όταν ξεπερνούν τα όρια του τι είναι επιτρεπτό. Τέλο πάντων, για την ένσταση αυτή, εάν, ξαναλέω, μπορούμε να την υποστηρίξουμε την ένσταση, θα μπορούσαμε μάλλον να την υποστηρίξουμε αν ήταν κατά τη αύξηση των μέγιστων επιτρεπωμένων ορίων των 3 μιλιγκράμμ. Αλλά επειδή δεν περιορίζεται σε αυτό, αλλά θέλει και να μειώσει τα όρια από τα, αυτά που ισχύουν τώρα. Αυτό το θεωρούμε επικίνδυνο. Διότι αυτό σημαίνει ότι η καλλιέργεια ελαιοδέντρων ιδίω στην Ιταλία, θα έχανε ένα σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία, τη φυτογενομική προστασία από την ξυλέλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η άρνηση να σκεφτούν ότι όπως και, όπως και άνθρωποι, τα φυτά έχουν προστασία, ανάγκη προστασίας στα φυτά η ιατρική ονομάζεται φυτογειονομική προστασία. Όταν εμεί είμαστε άρρωστοι ω άνθρωποι, πάμε σε ένα γιατρό. Δεν καταλαβαίνω γιατί ω άνθρωποι πρέπει να φροντίζουμε την υγεία μα ενώ στα φυτά απαγορεύεται. Επίση, μα λένε, ιδίω από την Ιταλική αντιπροσωπεία, ότι για να ε, αμφισβητηθεί το όριο αυτό που δεν υποστηρίζεται από όλε τι μελέτε, χρειάζεται τουλάχιστον ένα χρόνο συλλογή στοιχείων επιτόπου. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, δεν θα υποστηρίξω αυτή την ένσταση και καλώ του συναδέλφου να μην το κάνουν και να ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αύξηση μάλλον και ούτε να ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αύξηση των μέγιστων επιτρεπωμένων ορίων στα 3 μιλιγκράμμα ανά κιλό, να παραμείνουμε στα ισχύοντα και σήμερα, τα 0,9 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Εάν σκεφτούμε ότι χρειάζονται μειώσει, να περιμένουμε προηγουμένω να έχουμε συγκεντρώσει αρκετά επιστημονικά στοιχεία και να έχουν γίνει και δοκιμέ στην πράξη για να είμαστε βέβαιοι ότι κάτι τέτοιο έχει νόημα. Ιδάλω, ε, κάνουμε μια βουτιά στο κενό. Ευχαριστούμε κυρία Γκαρντίνη. Θα δούμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γνώμη έχει. Αλλά μην ξαναρχίσουμε τώρα το διάλογο και με τους ομιλητές για την ένσταση. Κυρία Ριβαζή, διότι είναι πολλοί συνυπογράφοντες. Αν όλοι θέλουν να δευτερολογήσουν θα γίνει. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απαντήσει. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε εσείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μιλήσει και να έχει τον τελευταίο λόγο. Αυτό που θέλετε να συζητηθεί μεταξύ σα μπορεί να το πει τώρα η Επιτροπή. Κυρία Γιούλικερ. Κύριε Γιούλικερ. Κυρία Γιούλικερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τη σημερινή συζήτηση. Έχουμε εδώ μια περίπτωση μάλλον σύγχυσης του ποιο είναι το νομικό πλαίσιο ποια είναι τα βήματα που έχουν γίνει και τι διασφαλίσεις έχουμε για να ορίζουμε μέγιστα επιτρεπόμενα όρια. Κάποιε αρχικέ παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα, ο κανονισμό για τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια που μα δίνει το πλαίσιο του στο οποίο εδώ αναλαμβάνουμε δράση έχει ω βασικό στόχο να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασία τη υγεία του καταναλωτή. Τα προτινόμενα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω είναι η πρόταση αυτή, έχουν πρώτα αξιολογηθεί με τεκμηριωμένα στοιχεία από την ΕΦΣΑ, με πολύ μεγάλη βάση δεδομένων και με σαφή επιβεβαίωση από την ΕΦΣΑ ότι όλα τα, όλες οι προτάσεις για τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια, τα MRL, είναι ασφαλείς, σωστές και σε τέτοιο επίπεδο που το επιτρέπουν τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει. Και συγκεκριμένα αυτό που έχουμε παρατηρήσει για τα ελαιόδεντρα και το επιτραπέζιο λάδι και ελιές. Εδώ λοιπόν η πρόταση ψηφίσματος δεν δικαιολογεί αυτή την μείωση σε 0,5 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Δεν βλέπουμε να υπάρχουν εδώ επιχειρήματα. Σκοπός του νομοθετήματος αυτού τη πρόταση για τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια ήταν κυρίω η προστασία του καταναλωτή. Δεν ήταν ε, σκοπό να ασχοληθούμε με την προστασία του περιβάλλοντο ή με του επικονιαστέ ή με την ε, υγεία των ζώων. Τα θέματα αυτά, και αυτή είναι η δεύτερη παρατηρήσή μου, καλύπτονται από ξεχωριστή ειδική νομική πρόταση και νομικό πλαίσιο. Αυτό αφορά την θέση στην αγορά των προϊόντων για την υγεία των φυτών τον ε, περίφημο κανονισμό του 07, 1107 του 2007. Εδώ υπάρχει και μια μελέτη αξιολόγηση κινδύνου που έγινε πρόσφατα και νομίζω ότι δεν τη λαμβάνει υπόψη η πρόταση ψηφίσματος εδώ η ένσταση. Αλλά και πάλι προσφάτως υπήρχε μια διεξοδική αξιολόγηση της ΕΦΣΑ που επιβεβαιώνει τα κριτήρια για την έγκριση της ακεταπριμίδης καλύπτονται και ότι δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία ούτε για τις μέλισσες και τους επικονιαστές. Διότι αυτό εξετάστηκε καταλεπτός και στις αρχές του 2018 η έγκριση της ακεταμιπρίδης ε, βρέθηκε ότι πληρεί τα κριτήρια για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και τους επικονιαστές. Οπότε ανανεώθηκε με, με στήριξη από τα κάτι μελη Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι το σύστημα, και νομίζω αυτό είναι και το πλεονέκτημα η δύναμή του είναι ότι κοιτάζει τα όρια ουσία αναουσία και όχι σε ομάδες ή σύνολα ουσιών όπως τα νεονικοτινοειδή. Έχουμε πιάσει την κάθε ουσία ξεχωριστά με δεδομένα, επιστημονικά στοιχεία, και πραγματικά είμαι βεβαία ότι έχει γίνει σωστά και στην περίπτωση της Ακεταμιπρίβης. Εάν λοιπόν με απασχολούσαν οι συνέπειε στο περιβάλλον ή επικονιαστέ στα πλαίσια του κανονισμού ε, MRL, θα ξεπερνούσε τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, διότι δεν καλύπτονται από αυτό το νομοθέτημα, αλλά από την ίδια την έγκριση της Ακεταμιπρίδης ήδη στις αρχές του 2018. Με αυτά κατανοεί, είναι σαφές ότι οι ανησυχίες που αναφέρει το σχέδιο ψηφίσματος, η ένσταση, δεν έχουν λόγο ύπαρξης, γιατί έχουν ήδη καλυφθεί στη διαδικασία έγκρισης της Ακεταμιπρίδης και μετά με την αναθεώρηση της διαδικασίας για τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια. Και ακόμα μια κουβέντα για τα προτιμνόμενα επίπεδα MRL, για τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα. Όπως είπα, η ΕΦΣΑ, και εδώ πιστεύω πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ως προς την αξιοπιστία της ΕΦΣΑ, διότι η ΕΦΣΑ είναι αξιόπιστος οργανισμός, έχουν επιβεβαιώσει ε, και διατρανώσει ότι είναι ασφαλείς αυτές οι ουσίες για τα ελαιόδεντρα, το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ηλιές και αν μιλήσουμε για την αύξηση που ζητάμε του μέγιστου επιτρεπόμενου οι καλές γεωργικές πρακτικές για να καταπολεμήσουμε αυτή τη μίγα των ελαιόδεντρων αυτό το έντομο που έχει καταστρέψει το ελεύθερα στην Νότια Ευρώπη, όχι μόνο η ξυλέλα, αλλά το ίδιο το ζωήφιο αυτό που δημιουργεί τρομερές ανησυχίες και μπορεί να εξαπλωθεί ευραίως. Βάσει λοιπόν όλων αυτών των δεδομένων, για το κατά πόσο είναι σωστά τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια, θεωρήσαμε ότι μπορούμε να τα αυξήσουμε ως εκεί. Υπάρχει επίσης και μια παρανόηση για το τι σημαίνει αυτό για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την προστασία των φυτών. Άκουσαν για τα, άκουσα για τα ταπλασιασμό των, της ποσότητας που χρησιμοποιούσαμε με τα προηγούμενα MRL. Δεν ε, το έχετε θέσει πολύ σωστά. Η αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου δεν έχει να κάνει πάρα πολύ με το βαθμό χρήσης των, ε, των φαρμάκων αυτών. Πρέπει να δούμε με προσοχή τους αριθμούς και το κατά πόσον ε, υπάρχει αύξηση όντω τριπλάσια, τετραπλάσια ή απλώς αυτό το 40% που θεωρούμε εμείς ότι είναι η πραγματικότητα. Πριν ολοκληρώσω, να πω ότι ο κανονισμός ως έχει είναι άκρο σημαντικός διότι αυτό που κάνει είναι ότι μειώνει τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια για πολλά ε, εμπορικά αγαθά όπως τα μήλα, τα ροδάκινα και, τα, ε, και γερμάδες. Και τα μέγιστα αυτά επιτρεπόμενα όρια πρέπει να αυξηθούν για να έχουμε καλύτερη προστασία της υγείας του καταναλωτή. Ξαναολοκληρώνοντας, να πω ότι είναι σημαντικός αυτός ο κανονισμός, ε, λαμβάνει υπόψη την ε, υγεία των καταναλωτών και είναι πλήρω ευθυγραμμισμένο με του στόχου του κανονισμού για τα μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξεπερνά τι αρμοδιότητες τη, ούτε ε, αγνοεί την ασφάλεια του περιβάλλοντο και την προστασία του, ούτε των μελισσών και των επικονιαστών. Αυτά τα έχουμε ήδη επιλύσει με την πρόσφατη αναθεώρηση του κανονισμού για τι δραστικέ ουσίε. Έτσι εγκρίθηκε η άδεια για την ακεταμιπρίβη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε λοιπόν, αλλά θα ψηφίσουμε έτσι κι αλλιώς αύριο. Και θα δούμε ποιο θα το... ποια θα είναι η έκβαση τη ψηφοφορία. Κλείνουμε το θέμα αυτό και περνάμε στο επόμενο. παράταση της περίοδου έγκρισης για διάφορες δραστικές ουσίες, όπως το κλωροπυρηφός. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή. Η κυρία Γιούλικερ, εάν θέλει να μας παρουσιάσει αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Η ουσία αυτή κλορπυριφός και το κλωρπυριφός μεθύλ εγκρίθηκαν το 2006 μετά από μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Η έγκριση αυτών των δραστικών ουσιών επανεξετάζεται για να διαπιστώσουμε εάν μπορούμε να ανανεώσουμε ή όχι την έγκριση. Η οι ισχύουσες εγκρίσεις ε, λήγουν το 2020 τον Ιανουάριο και πρόσφατα παρατάθηκαν με την υποστήριξη των κρατών μελών. Τον Οκτώβριο συγκεκριμένα το 2018 για να επιτραπεί η ολοκλήρωση της ε, αναθεώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού περί φυτοφαρμάκων 11 ε, ε, του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να παρατείνει τη χρήση δραστικών ουσιών όταν για λόγους που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του ετούντος ε, μπορεί να λήξει η έγκριση πριν από την ανανέωση απόφασης. Και ήταν νομικό το κείμενο που παρέθεσα, ζητώ συγγνώμη, αλλά εάν υπάρχουν αιτίε ε, που δεν οφείλονται σε λάθο πράξη του ετούντο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να παρατείνει την έγκριση. Και αυτό λοιπόν ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε και αυτό κάναμε. Η έκθεση αξιολόγηση του ε, σχετικού κράτους μέλους ε, της Ισπανίας, δηλαδή έχει καθυστερήσει λόγω της πολυπλοκότητας των τεχνικών πληροφοριών που πρέπει να αξιολογηθούν. Να είμαστε λοιπόν απόλυτα σαφείς, ε, συνεχίζεται η επανεξέταση και ευθυγραμμιζόμαστε απόλυτα με την νομοθεσία. Δηλαδή παρατείνουμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα την έγκριση για να επιτρέψουμε την ολοκλήρωση της έκθεσης. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και πραγματοποιείται με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά και ε, τεχνολογικά στοιχεία εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη συμμετέχουν, όπως και η ΕΦΣΑ. Όταν ολοκληρωθεί η επιστημονική αξιολόγηση, η ΕΦΣΑ θα δημοσιεύσει τα συμπεράσματά της, τα οποία περιμένουμε το δεύτερο εξάμεινο του 2019 και που θα βασίζονται σε ανάλυση και μάλλον με βάση αυτή την ανάλυση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει εάν θα προτείνει ανανέωση της έγκρισης ή θα επιλέξει άλλη πορεία. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι τα προηγούμενα έτη που μιλούσαμε για μέγιστα επίπεδα ε, καταλήπων, ε, τα επίπεδα για το κλωρπυρηφός μετά από εκτενείς έρευνες το 2015 και το 2017 ε, προσαρμόστηκαν. Εάν χρειαστεί περαιτέρω δράση πάνω στα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια καταλήπων, ε, ε, θα σας ενημερώσουμε. Είχαμε πρόσφατα αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα ήθελα να τονίσω ότι οι αξιολογητές εξετάζουν τα δεδομένα αυτά καθεαυτά, όχι απλά τη σύνοψη που δίδεται. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι σε αντίθεση με όσα έχουν αναφερθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι προσιλωμένη στον στόχο ε, απαγόρευσης στην αγορά επικίνδυνων ουσιών. Ουσιών δηλαδή που δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρίβαζη, παρακαλώ. Από πλευράς Επιτροπής νομίζω ότι δεν βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Εμάς μας ενδιαφέρει η προστασία των καταναλωτών και έχουμε να κάνουμε με ένα όργανο που θεωρείται μερόληπτο. Αν κάποιος αμφισβητεί αυτό, ε, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλιώς δεν θα υπήρχε ένσταση, όπως καταλαβαίνετε. Εσείς θεωρείτε ότι είναι τέλεια εμείς όχι. Λοιπόν, με εκπλήσουν κάπως αυτά που λέτε. Γιατί το όσο ξέρουμε ότι είναι τοξικό, ότι έχει φόσφορο, ότι χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα πέντε παρασιτοκτόνα που περισσότερο εντοπίζεται μέσα στα ποροκυπευτικά που καταναλώνουμε και έχει υπάρξει έτοιμα για επαναδιαδότηση. Η Ισπανία δεν έχει δώσει τα δικά της ε, τεκμήρια. Γιατί έκανε τόσο καιρό να αξιολογήσει αυτό το παρασιτοκτόνο. Και εφόσον ο ετών η χώρα μέλος μάλλον καθυστερεί τόσο πολύ, εσείς λέτε καλά. Και θα σας δώσω μια λεπτομέρεια εδώ, γιατί υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα με το παρασιτοκτόνο αυτό. Πρώτα απ' όλα, δεν επιτρέπεται πια σε 8 ευρωπαϊκές χώρες. Δανία, Φιλανδία, Γερμανία, Ελλανδία, Λετωνία, Λιθουανία, Σλοβενία και Σουηδία. Και γιατί το έχουν απαγορεύσει αυτές οι χώρες? Γιατί έχουν τα δεδομένα. Γιατί έγιναν διάφορες ανεξάρτητες μελέτες που έδειξαν ότι πρόκειται για ένα παρασιτοκτόνο το οποίο είναι νευροτοξικό, ε, πρόκειται για ενδοκρινικό διαταράκτη κλπ. Και, Και γι' αυτό το απαγορεύσανε. Και εμεί κάναμε μια δοκιμή στα μαλλιά. Αναλύσαμε 150 ε, πειράματα κάναμε σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, αναλύοντας ε, τις τρίχες των ανθρώπων και στη Γερμανία που απαγόρευσε αυτό το παρεστοκτόνο. Ε, λοιπόν, ακόμα το βρίσκουμε στα μαλλιά μας. Ακόμα δηλαδή και αν έχει απαγορευτεί ένα παρεστοκτόνο, παρόλα αυτά οι ίχνοι του εξακολουθούν να βρίσκονται στις τρίχες. Και αυτό τι σημαίνει ότι παραμένει ένα μήνα, γιατί θέλει ένα μήνα η τρίχα για να μακρύνει ένα εκατοστό. Οπότε, εμείς σας ζητούμε με όλες τις πανεπιστημιακές μελέτες που έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα που δείχνουν ότι αυτά που λένε οι βιομηχανοί ελαχιστοποιούν την αξιολόγηση κινδύνου. Και επίσης έχουν γίνει μελέτες, έτσι. Σε σχέση με αυτή την επιστημονική αμφιβολία ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορεύσει αυτό το παρασιτοκτόνο. Μα κοιτάξτε τι γίνεται με τους καταναλωτές. Κανείς δεν θέλει πια προϊόντα που οδηγούν σε νευροτοξικά προβλήματα, απώλεια διανοητικών ικανοτήτων κτλ. Ενώ εσείς τι κάνετε, το παρατείνετε άλλο ένα χρόνο. Και ελαχιστοποιείτε την αξιολόγηση κινδύνου. Πριν δεν μπόρεσα να σας απαντήσω, αλλά όταν μειώσαμε το MLR για το προηγούμενο παρασιτοκτόνο, το κάναμε για το προκυπευτικά, γιατί καταλάβαμε ότι είναι επικίνδυνο και ότι πρέπει να έχουμε όσο γίνεται λιγότερα κατάλοιπα. Αλλά δεν θέλουμε να το κάνουμε με την ελιά και το λεόλαδο. Υπάρχει πρόβλημα εφόσον μειώνουμε τις οριακές τιμές στο προκυπευτικά. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω καθόλου. Εσείς στο μυαλό σας δεν έχετε καθόλου την προστασία του καταναλωτή. Και σας λέω, Επιτροπή, έχουμε ευρωεκλογέ του χρόνου. Εμείς πάντα επειδή ακριβώς είμαστε υπέρ της Ευρώπης, λέμε πάντα ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύει. Όμως με τη λειτουργία της ΕΦΣΑ εσείς καταστρέφετε αυτήν την φυτογενομική προστασία που σιγά σιγά φτιάξαμε εδώ στην Ευρώπη και είσαστε συνένοχοι του λαϊκισμού που κινδυνεύει να υπερισχύσει στην Ευρώπη. Πρέπει να το απαγορεύσετε αυτό βάσει της αρχής της προφύλαξης. Κοιτάξτε όλες τις ε, μελέτες που έχουμε σήμερα και θα το απαγορεύσετε. Ενώ εδώ έχουμε την αίσθητη ότι είσαστε υπέρ των μεγάλων βιομηχανιών ε, που παράγουν ε, αυτά, αυτές τις ουσίες, τις δραστικές ουσίες των παρασιτοκτόνων. Είσαστε συνένοχοι. Όταν λέτε ότι συμφωνούν οι χώρε μέλη, δεν είναι αλήθεια. Οχτώ χώρε το έχουν απαγορεύσει αυτό το παρασιτοκτόνο. Άρα δεν ισχύει αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε κυρία Ριβαζή. Ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω 100% με αυτά που μόλις είπε η κυρία Ρίβαζη. Ειλικρινά, από τότε έχω έρθει εδώ. Είναι ε, ίσως η πρώτη και τελευταία θητεία για μένα, βεβαίως. Ε, δεν έχω δει ποτέ να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης. Αυτό που θεωρείται εδώ το καμάρι των ευρωπαϊκών θεσμών δεν το έχω δει ποτέ να εφαρμόζεται. Και κάθε φορά που αρχίζει μια καινούργια συζήτηση, ξανανοίγει μια παλιά συζήτηση για το ποιε είναι οι προθεσμίε εκπνοή των ε, προηγούμενων εγκρίσεων, όλο κάτι γίνεται. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα φετοφαρμακό το οποίο έχει νευρολογικέ επιπτώσει στην υγεία των υπείων, των βρεφών. Και το λέει ε, επιστημονική κοινότητα από τι ε, πλέον έγκυρε που υπάρχουν, ε, η Insta, ε, για την ε, ενδοκρινολογική, ως ενδοκρινολογικός καταρα... έχει, έχει εντοπιστεί επίση και ως ε, καρκινογόνο ουσία και με πάρα πολλέ σορευμένε επιπτώσει για το περιβάλλον. Ωστόσο, η ΕΦΣΑ, που είναι η μόνη αρχή που είναι τυπική κα εγκεκριμένη για να ε, τοποθετηθεί και να εκδώσει μια, ένα επιστημονικό πόρισμα δεν καταφέρει να επηρεάσει καν την Επιτροπή, απλώς αποφασίζει να παρατείνει την έγκριση. Για κάθε λοιπόν διαδικασία διοδότηση για την ουσία αυτή που είναι επικίνδυνη και για κάθε επίπτωση που βλέπουμε να υπάρχει στου πολίτες που είναι επιζήμια, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν θα κάνω καν ερώτηση, απλώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρω ότι θα απαντήσει. Οι πολίτε που θα ακούσουν αυτή την παρέμβαση, ίσω να σκεφτούν ότι με την μπανάνα και τα πλαστικά που την περιβάλλουν ή το άλλο επικίνδυνο χημικό που χρησιμοποιείται στα ε, πλαστικά ε, θα το πάρουν χαμπάρι και με όλα αυτά έχω να σας ευχηθώ καλή όρεξη. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Η κυρία Γιούλικερ πάλι. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για τις παρεμβάσεις. Πρέπει νομίζω να σας πω δύο πραγματάκια. Δεν υποβαθμίζω καθόλου τους κινδύνους. Απλώς σας λέω η ουσία αυτή εξετάζεται, είναι υπό εξέταση και ευχαρίστως μόλις έχουμε τη διαδικασία αυτή ολοκληρωμένη, να έρθω με το πόρισμα να σα το παρουσιάσω και να αναλάβουμε τη σχετική δράση. Δεν υποβαθμίσω κανένα κίνδυνο. Ούτε έχω καμία διάθεση, ούτε η Επιτροπή έχει καμία ε, πρόθεση, ούτε η ΕΦΣΑ, να καταστρέψουμε την προστασία των καταναλωτών. Αυτό είναι μάλλον κάτι το οποίο θα το αντέκροα με στεναρότητα. Και από την άλλη υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Η αρχή της προφύλαξης αναφέρθηκε και χρησιμοποιείται και έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένος και να σας θυμίσω το αποτέλεσμα του γενικού μας νόμου για τα τρόφιμα το χρησιμοποίησαμε για την βισφενόλη α αν το θυμάστε Αλλά, όπως είπα, περιμένουμε την έκβαση αυτής της διαδικασίας, η οποία θα μας δώσει τη βάση για να προχωρήσουμε στις απαραίτητες κινήσεις. Κυρία Ριβαζή, είπατε ότι η ουσία αυτή απαγορεύεται σε ένα-δυο μελη Οκτώ. Νομίζω σωστότερη θα ήταν ε, η διατύπωση τα προϊόντα προστασίας των φυτών δεν επιτρέπονται σε κάποια κράτη-μέλη. Όντως, αυτό είναι φυσιολογικό. Διότι αν δεν υπάρχει κάποιο ζυζάνιο ή κάποιο άλλο ζωήθιο που να απειλεί τα φυτά, δεν έχει λόγο να δώσει άδεια το κράτος μέλος ε, στα συγκεκριμένα προϊόντα, ακόμη και αν επιτρέπονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό ισχύει για ένα σωρό δραστικέ ουσίε. Εάν λοιπόν μπορούσα να ολοκληρώσω, τι θα έλεγα. Οπωσδήποτε, μόλις εκδοθεί η σχετική γνωμοδότηση, θα αναλάβουμε δράση. Είναι σαφές. Και επίσης, σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζουμε τους κινδύνους. Είμαι βεβαίω ότι αυτό που προτείνουν οι αξιότιμοι κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές ε, θα ε, αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης κινδύνου από τα κράτη-μέλη και τους επευθύνους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ΕΨΑ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ε, έτσι κλείνουμε τη συνεδρίασή μας. Θα σας δω αύριο το πρωί για τις ψηφοφορίες στις 9. Καλό βράδυ.